Ε, good morning. Καλημέρα. Έχουμε κάποιους προσκεκλημένους για να ανταλλάξουμε απόψεις ε, And, ε, we are missing... για την uh, πολιτική συνοχή μετά το 2013. Ε, κάποιος είναι ακόμα στην προσπαθεί να πάρει το πάσο του για να μπει. Ε, ας ακούσουμε λοιπόν τώρα την κυρία Αν Σοφή Παράν από την Age Platform Europe. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσω με λίγα λόγια για την οργάνωσή μου για να καταλάβετε ε, τι θα πω. Το AIDS είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που ενώνει πάνω από 2 εκατομμύρια ηλικιωμένους στην Ευρώπη από 30 χώρε κρατη με ηλικία υποψηφίε χώρε και στόχο έχουμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των ηλικιωμένων στη λήψη αποφάσεων. Δηλαδή μιλάμε για τους άνω των 50 το 1 τρίτο του πληθυσμού, 150 εκατομμύρια. Το πώς το προσεγγίζουμε δεν είναι μόνο μέσω της πρόωθησης των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους, αλλά παίρνουμε μια προσέγγιση συνολική για ολόκληρη τη ζωή, δηλαδή λύσεις που είναι καλές και για τους ηλικιωμένους αλλά και για τις άλλες γενιές, ειδικά τις νεότερες γενιές που πιέζονται αυτή τη στιγμή. Αυτό σας δίνει μια ιδέα της προσέγγισής μας ε, που, είναι, που προωθούμε με ομοφωνία στο δίκτυό μας. Δεν θα μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, ξέρω πώς διαπραγματεύεστε, έχετε κάνει προτάσεις και θα έλεγα πως στηρίζουμε αυτά τα οποία λέτε, την προσέγγισή σας και κάτι το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι το εξής. Ε, πρέπει να στηρίξουμε και να προωθήσουμε μια καλύτερη επίπεδη διακυβέρνηση. Συνεργαζόμαστε με τοπικές και περιφερειακές αρχές στο πλαίσιο της καμπάνιας μας για ε, ένα περιβάλλον φιλικό προς ηλικιωμένους. Τι εννοούμε δηλαδή, είπε φιλικό προς όλες τις ηλικίε. Και εκεί θα θέλαμε βεβαίω πολύ καλύτερη συνεργασία και ευκαιρία συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της διακυβέρνησης. Γιατί μας λένε οι τοπικές αρχές πως προσπαθούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πληθυσμών κοιτώντας βεβαίως τις διάφορες ε, ηλικιακέ ομάδες αλλά εάν δεν τις υποστηρίζει η περιφέρεια, εάν υπάρχει η περιφέρεια ε, και το εθνικό επίπεδο δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, ε, οργάνωσε πέρσι τον Ιούνιο μια σχετική διάσκεψη και εκεί πέρα φάνηκε πως οι χώρες οι οποίες έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα είναι οι χώρες οι οποίες ε, έχουν καλή συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης, δηλαδή συμφωνούν ότι έχουν μια πρόκληση, όπως η δημογραφική αλλαγή μαζί με την κλιματική αλλαγή. Οι χώρες οι οποίες μπόρεσαν λοιπόν να προωθήσουν μια καλή συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων ε, διακυβέρνησης είναι αυτές οι οποίες έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Για μας λοιπόν αυτή η προσέγγιση είναι κάτι το οποίο ελπίζουμε πως θα υποστηριχθεί από την πολιτική συνοχής και τα μέσα χρηματοδότησης. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Καινοτομίας για την Υγιή που είναι ένα νέο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων μεταξύ αρχών αλλά και του κλάδου ερευνητών και γενικώ της κοινωνίας των πολιτών. Έχουμε λοιπόν μια εκστρατεία για να προωθήσουμε ακριβώς το περιβάλλον, το φιλικό προς τη γύρανση ε, την ευρεία έννοια και κάτι το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο δημάρχων και περιφερειακών αρχών για τη δημογραφική ε, αλλαγή ή τα, το περιβάλλον το φιλικό προς τη Δεν ξέρουμε ακόμα ποιος θα είναι ο τίτλος. Γιατί το κάνουμε αυτό. Πρώτα απ' όλα έχουμε την ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών του Μαΐου που μας πέρασε που επίσης ζητάει μια ανταπόκριση στη δημογραφική αλλαγή ως μια βασική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές. Αλλά αυτό δεν αντικατοπτρίζεται πάντα στις ε, προτεραιότητες των εθνικών αποφάσεων. Έχω δει κάποιες τροπολογίες λοιπόν οι οποίες πραγματικά τονίζουν περισσότερο την ανάγκη να ενσωματωθεί αυτή η πρόκληση. Οπότε για εμάς αυτό είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε να στηρίξουμε Να προσπαθήσουμε δηλαδή να δούμε αν μπορούμε να ενισχύσουμε την ε, έμφαση για την ε, στην προσέγγιση για τον κύκλο ζωή, θα έχετε ακούσει τι σχετικέ γειτονιέ, παραδείγματο χάρη. Περισσότερε τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ πρέπει να συμφιλιώσουν ανάγκε οι οποίε φαίνονται κάπω διαφορετικέ ε, εκ πρώτη όψεω, αλλά εντό του συμφώνου θα θέλαμε επίση να εισεχθεί η διάσταση τη καινοτομία κάτι το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο και πρέπει να ενισχυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίσης η σύνδεση με την περιβαλλοντική διάσταση. Κατόπιν υπάρχει μια τροπολογία για τη ΦΕΝΤΕΡ για να επιτραπεί η χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία. Ειδικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις περιφέρειες που χρειάζεται ε, να επενδύσουν περισσότερο για να γίνουν πιο φιλικό προς όλες τις ηλικίε ε, το περιβάλλον τους. Όλες τις ηλικίε, όχι μόνο, όπως είπα, τις ε, πιο μεγάλες. Αυτά ήθελα να τονίσω αυτή τη στιγμή. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα για τις συγκεκριμένες τροπολογίες που έχετε προτείνει. Αν το θεωρείτε χρήσιμο να σας στείλουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τροπολογίες, Ευχαριστώ μπορούμε να σας στείλουμε αργότερα. Ήμασταν πάρα πολύ, πολύ άσχολοι με το ευρωπαϊκό έτος ε, ενεργούς ε, γύρανσης ε, και τρέχουμε πανικόβλητοι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για μας και ελπίζουμε οι κανόνες να βελτιωθούν για να φροντίσουμε τα μέσα αυτά βέβαια να έχουν και το καλύτερο αποτέλεσμα δίνοντας την δυνατότητα στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο να εκδιπλώσει το δυναμικό του, με τη στήριξη βεβαίως του εθνικού επίπεδου διοίκησης, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει και κάποιος λόγος για το τι θα χρηματοδοτηθεί αργότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Παράου. Θα δώσω λόγο στον κύριο Ζιλιέν Ντιγιόλ που εκπροσωπεί το Housing Europe. Thank um, Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Στην παρουσίασή μου θα ασχοληθώ με τρία στοιχεία. Καταρχάς θα μιλήσουμε για την θεματική συγκέντρωση όσον αφορά την στέγαση χαμηλού κόστους και αναφέρομαι εδώ πέρα στο άρθρο 4 της του σχετικού κανονισμού θα αναφερθώ επίσης στην ε, δυνατότητα μέσω της στέγασης να αντιμετωπίσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό και αναφέρομαι εδώ πέρα στο άρθρο 5 του κανονισμού και στη συνέχεια την ε, δυνατότητα μεγαλύτερης ε, ενσωμάτωσης της κοινωνίας καθώς επίσης και μελλοντικών επενδύσεων μπορεί να γίνουν και ολοκληρώνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στην καταμέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου που μπορεί να έχουν αυτές οι επενδύσεις. Και όλα αυτά θα γίνουν από την σκοπιά, την οπτική γωνία της ε, φτηνής στέγασης. Εκπροσωπώ την Housing Europe Federation, την ε, Ομοσπονδία Οργανώσεων Κοινωνικής Στέγασης στην Ευρώπη. Καταρχάς, για ποιο λόγο είμαστε υπέρ της ε, θεματικής συγκέντρωσης όσον αφορά την κοινωνική στέγαση. Για δύο λόγους καταρχάς. Πρώτον, όπως βλέπετε και στην οθόνη, υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά το ζήτημα της ενέργειας, της χρησιμοποίησης ενέργειας από τους Ευρωπαίους πολίτες. Είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας κοινό ορισμός όσον αφορά την λεγόμενη ενεργειακή ένδυα στην Ευρώπη, προκειμένου να υπάρχουν και σχετικές πολιτικές καταπολέμησής της. Έχουμε αριθμητικά δεδομένα και από τη Eurostat, όπου φαίνεται ότι τουλάχιστον 52 εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να ζεστάνουν επαρκώς το σπίτι τους. Θεωρούμε λοιπόν ότι πλήττονται από την ενεργειακή αυτή ένδυα, από την ένδυα καυσίμων. Δεν έχουν τα χρήματα για να αγοράσουν καύσιμα. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί δείκτες που χρησιμοποιούν και πραγματικά υποστηρίζουν αυτή τη διαπίστωση. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο είμαστε υπέρ της θεματικής συγκέντρωσης με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα είναι γιατί ε, πιστεύουμε ότι πραγματικά θα μπορούσαν να γίνουν οι σχετικές επενδύσεις όσον αφορά τις στεγαστικές δαπάνες και ξέρετε ότι υπάρχουν ήδη κάποιες μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχουν πολύ θετικές μακρο, μακροοικονομικές επιπτώσεις από τη χρησιμοποίηση της οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στον τομέα της στέγασης. Επίσης υπάρχει μια άλλη αντίδραση όσον αφορά το ζήτημα της απασχόλησης. Ξέρετε ότι ε, το να έχουμε κτίρια τα οποία θα είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον μπορεί σε κάποιους τομείς να οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας, αλλά κυρίως να οδηγήσει σε δημιουργία θέσεων εργασίας. Πολύ περισσότερες είναι θέσεις εργασίας από αυτές που θα χαθούν. Αν συγκρίνουμε τα στοιχεία αυτά με τις ανάγκες σε επενδύσεις, 60 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2020 αναέτος, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και αν συνδυάσουμε τα στοιχεία αυτά με την οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα, βλέπετε πραγματικά ότι η κατάσταση πιέζει ιδιαίτερα και γι' αυτό το λόγο εμείς είμαστε υπέρ μιας φιλόδοξης χρηματοδότησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι οι περιφέρειες θα είναι υποχρεωμένες να δαπανίσουν χρήματα για τη στέγαση. Εμείς πάντως πιστεύουμε ότι η στέγαση θα είναι η πρώτη επιλογή όσον αφορά τις πολιτικές οικονομικής αποδοτικότητας. Δεύτερον τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν συγκεκριμένε επενδύσει κατά προτεραιότητα. αναφέρουμε εδώ πέρα στο άρθρο 5 του Κανονισμού Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακή Ανάπτυξη. Πολλά εμπλεκόμενα μέρη κάνανε διάφορε προτάσει όσον αφορά τι προτάσεις που θα πρέπει να γίνουν για τις επενδύσεις. Εμείς θεωρούμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υποστηρίζεται από το Κοινοβούλιο είναι καλή, είναι συνεκτική. Αν δούμε το ζήτημα της στέγασης, βλέπετε εδώ πέρα ότι υπάρχουν διαφορετικές εναλλακτικέ λύσεις όσον αφορά τις, ε, την κοινωνική στέγαση, όσον αφορά τα φιλικά προς το περιβάλλον σπίτια, όσον αφορά την ε, στέγαση η οποία θα είναι φιλική προς το περιβάλλον. Και η Αν Σοφία αναφέρθηκε σε κάτι το οποίο έχει εισάγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τροπολογία για την παράγραφο 9 του άρθρου 5, όπου προβλέπεται ότι κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα μπορούν να αφιερωθούν περισσότερο στη σωστή ανάπτυξη και αναγέννηση των πόλεων. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά σχέδια αυτή τη στιγμή τόπου, πάρα πολλά προγράμματα και δεν είναι δυνατόν όλα αυτά τα σχέδια, όλα αυτά τα προγράμματα να συνδυαστούν και να χρηματοδοτηθούν. Αν θέλουμε λοιπόν να επικεντρωθούμε στις επενδύσεις προς την κοινωνική στέγαση, προς τις κοινωνικές υποδομές, θεωρώ ότι μπορούμε όντω να χρησιμοποιήσουμε τα προγράμματα αυτά και αξίζει αν θέλουμε πραγματικά να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, τη φτώχεια με συγχωρείτε και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αν δούμε εδώ πέρα το συνολικό εισόδημα των οικοκυριών που ζουν σε εργατικές κατοικίες στη Γαλλία, βλέπετε ότι το 2006 τα άτομα τα οποία βρίσκονται εδώ πέρα στο πρώτο τεταρτημόριο αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων εργατικών κατοικιών. Αν πραγματικά λοιπόν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, θα πρέπει να ασχοληθούμε το ζήτημα της κοινωνικής στέγασης. Βλέπετε λοιπόν ότι ένας πολύ λογικός τρόπος να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους της ε, Ευρώπης 2020, μάλλον ένα από τους στόχους, τη μείωση της φτώχειας στην Ευρώπη. Τέλος. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάρα πολλά εργαλεία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Έχουμε εδώ πέρα δύο πολύ σημαντικά σημεία αναγνωρίζουμε ότι όλε οι πολιτικέ περιφερειακή ανάπτυξη χρειάζονται μια ολοκληρωμένη δράση. Αυτό ισχύει για την πολιτική για τι κλιματικέ αλλαγέ και βλέπουμε εδώ πέρα ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα για το πώ μπορεί να συνδυαστεί η πολιτική αυτή τη κοινωνική στέγαση με την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών σε τοπικό επίπεδο. Ισχύει όμω η διασύνδεση αυτή και για τι κοινωνικέ πολιτικέ. Αν θέλουμε, για παράδειγμα, να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της ε, ροής των κεφαλαίων και την καταπολέμηση της φτώχειας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς τα τοπικά αυτά δίκτυα και τα προγράμματα κοινωνικής στέγασης. Κάτι ε, ενδιαφέρον για την ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση των τοπικών εργαλείων είναι το ότι ε, αναγνωρίζεται πάρα πολύ η συμμετοχή, η συμβολή των χρηστών. Εδώ πέρα όμως υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Αναφερόμαστε λοιπόν εμείς εδώ στο άρθρο 28 έως 32 του σχεδίου κανονισμού, καθώς επίσης και για το άρθρο που έχει να κάνει με το ITI και υποστηρίζουμε επίσης τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενδυναμώνουν το ρόλο των εταίρων σε όλες τις αποφάσεις ακόμα και στην επιλογή των κριτηρίων για τη στρατηγική. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηριζόταν μάλλον πάρα πολύ στο ρόλο των κρατών μελών. Εμεί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να αποφύγουμε να μην εμπλακούν όσο θα έπρεπε οι α, τοπικοί εταίροι. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι τοπικοί εμπλεκόμενοι να μπορούν και αυτοί να καθορίζουν ποια είναι τα κριτήρια για τη στρατηγική που ακολουθούμε. Θα σας δώσω τώρα δύο παραδείγματα για το πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε περισσότερο τις τοπικές ομάδες κοινωνικής ενσωμάτωσης και πώς μπορούμε να εμπλέξουμε, εμπλέξουμε περισσότερο το ITI στα προγράμματα αυτά τα οποία προωθούμε. Κυρίως στα προγράμματα κοινωνικής στέγασης και θεωρούμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης αλλά και από άλλα ταμεία. Η Anne-Sophie Paron αναφέρθηκε σε ένα πρόγραμμα το οποίο αναφέρεται στις γειτονιές, πώς μπορούμε δηλαδή να έχουμε ολοκληρωμένες οντότητες στα πλαίσια των διαφόρων γειτονιών. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις θεωρούμε ότι οι τοπικές αυτές ομάδες μπορούν να δραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ένα σημαντικότερο ερώτημα, και όχι μόνο για το ελεγκτικό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πιστεύουμε πραγματικά ότι μπορούν να συμβούν κάποιες βελτιώσεις και χρειάζεται πραγματικά η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το πρώτο σκέλος του ερωτήματο, εμεί θεωρούμε ότι όντως η ε, μέτρηση, η καταμέτρηση μάλλον υπολογισμός ε, των κοινωνικών επιπτώσεων, του κοινωνικού αντικτύπου της πολιτικής αυτής ε, είναι πολύπλοκος. Θα πρέπει πολλές φορές να χρησιμοποιούμε διάφορες παραμέτρους, ακόμα και την παράμετρο του κόστους. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να βασιστούμε αυτή τη στιγμή στην πρόοδο που είχε σημειωθεί εξαιτία τη δραστηριοποίηση πολλών τοπικών φορέων, ιδίω στο ζήτημα τη κοινωνική στέγασης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένας περιορισμένος αριθμός δικτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί που θα συμπληρώνεται από δείκτες οι οποίοι θα δημιουργούνται επί τόπου από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Δεν μπορούμε να έχουμε μόνο μία και μοναδική ομάδα δικτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα είναι πραγματικά σε θέση να καταμετρούν τον κοινωνικό αντίκτυπο. Ζήτημα ιδιαίτερα πολύπλοκο όπως σας είπα. Δεύτερο τώρα σκέλος του ερωτήματος απαιτείται η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς βασιζόμενοι στην εμπειρία που έχουμε με διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορες μελέτες, μπορούμε να πούμε ότι ε, τουλάχιστον όσον αφορά τα διατροτικά ταμεία και τη χρησιμοποίησή τους, πραγματικά βελτιώθηκε πάρα πολύ η συμβολή του στη δημιουργία των ε, προγραμμάτων κοινωνική στέγαση και ενίσχυσαν πάρα πολύ τα κονδύλια αυτά του τοπικού φορεί. Αυτό μόνο αποτελεί μια καταπληκτική απόδειξη τη ε, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Χωρί τα τρωτικά ταμεία και χωρί τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη, πάρα πολλά προγράμματα δεν θα είχαν δει το φω τη ημέρα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα και είμαι στην ε, διάθεσή σας για να σας βοηθήσω και εγώ με όλες τις διαπραγματεύσει τις οποίες διεξάγετε. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. you, Ευχαριστούμε κύριε Γκίγιο. Ο κύριος Σεμπαστιάν Κοντινό από το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση έχει το λόγο τώρα. Γεια σας. Το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση εργάζεται εδώ και 10 χρόνια για την πολιτική συνοχής. Θα ήθελα να τονίσω τέσσερα θέματα προτεραιότητες που συνιστούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλα, θα μιλήσω εξ ονόματος επτά μη κυβερνητικών οργανώσεων που διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο και εργάζονται και στις Βρυξέλλες και στις περισσότερες χώρες μέλη για την προσοχή του περιβάλλοντος. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη συνεκτικότητα μεταξύ των στόχων, των προτεραιοτήτων και της συνοχής, ώστε να δημιουργήσουμε καταστάσεις επικεδής για όλους, να βελτιωθεί η ευημερία των πολιτών, προστατευτεί τον περιβάλλον και να υλοποιηθούν οι στόχοι της Ευρώπης 2020. Οι τέσσερι τομείς κλειδιά που θα ήθελα να τονίσω σήμερα είναι οι εξής. Πρώτα απ' όλα, οι δύο αφορούν την σωστή πολιτική και δεύτερον, τον σωστό τρόπο εφαρμογής πολιτικής συνοχής. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να γίνει σωστή εκτίμηση σχεδίων και προγραμμάτων με την προστασία του περιβάλλοντος. Δεύτερον, να χρησιμοποιούνται αποδοτικά οι, ενέργεια, οι πηγές ενέργειας που έχουμε και για την προστασία του οικοσυστήματος και ό,τι κάνουμε στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής να είναι πιο ορατό και για το στάδιο εφαρμογής θα πρέπει να γίνει η σωστή εφαρμογή. Τι σημαίνει αυτό. Τα αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής που θα εφαρμόσουμε να βασίζονται σε σωστά κριτήρια τα οποία θα καθορίσουμε εκ των προτέρων ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά την πολιτική μας. Το δεύτερο θέμα που αφορά την εφαρμογή της πολιτικής είναι να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε πάρα πολύ δυνατές ε, ε, εταιρικές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα, σε διακυβερνητικό και σε όλα τα άλλα και να έχουμε το σωστό τρόπο εφαρμογής όλων αυτών των έργων. Και βεβαίω εδώ επίσης έρχεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε εργαστεί για αυτό το θέμα ε, βάσει διάφορων κανονισμών. Το πρώτο το οποίο υποστηρίζουμε είναι ότι η βιοπικιλότητα θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο να εμφανίζεται περισσότερο και να είναι πιο ρητά επεκφρασμένο στα πλαίσια της ε, πολιτικής ε, τις οποίες θέλουμε να κάνουμε για την προστασία των οικοσυστημάτων, εάν αυτό δεν αναφέρεται ρητός και με σαφή τρόπο στους κανονισμούς, κανείς δεν θέλει να υλοποιήσει τους στόχους. Δεύτερον, οι διατάξεις που αφορούν την, προστασία του, την κλιματική προστασία. Θα έπρεπε στο άρθρο 48 για την εκτίμηση των προγραμμάτων να γίνεται η, σωστό, η σωστή εκτίμηση των επιπτώσεων ε, των κλιματικών αλλαγών στην προστασία του περιβάλλοντος. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ο ρόλος σας είναι πάρα πολύ σημαντικός για να γίνει αξιολόγηση των προγραμμάτων και να δίδεται καλύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτύσσονται σχέδια και προγράμματα τα οποία δεν θα είναι δαπανηρά και ανετικά. Τελευταίο βασικό στοιχείο κατά την άποψή μας στις κοινέ διατάξεις είναι η αρχή των εταιρικών σχέσεων. Πρόκειται για ένα λεπτό θέμα με το Συμβούλιο. Ξέρουμε ότι γίνεται προσπάθεια στο θέμα αυτό να ασκηθεί πίεση στα κράτη-μέλη, διότι επιτόπου οι συνάδελφοι ξέρουν πόσο δύσκολο είναι να εμπλακεί κανείς στον σχεδιασμό των προγραμμάτων και δημοσιοποίησαμε μία κοινή επιστολή 42 θεσμικών οργάνων οργανώσεων της Κοινής των πολιτών ε, ομοσπονδιών όπως αυτή τη των μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων ενώσεων όπου όλοι εκφράζουν την αρχή ε, της ε, σωστής εταιρική σχέση, η οποία πρέπει να υπάρξει σε κοινοτικό επίπεδο. Ελπίζουμε ότι εσείς δεν θα υποχωρήσετε μπροστά στις θέσεις του Συμβουλίου που προσπαθεί να αποδυναμώσει αυτή την αρχή. Πιστεύουμε ότι η αρχή της εταιρικής σχέσης είναι πρωταρχή σημασία για να μπορέσουμε να έχουμε μία καλύτερη εφαρμογή της πολιτικής συλλογή σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο και έτσι θα κάνουν την πολιτική συνοχή πιο αποδοτική κυρίως την ε, εποχή αυτή των οικονομικών δυσκολιών. Τώρα, όσον αφορά τον κανονισμό που αφορά το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το μεγάλο θέμα αφορά την ενέργεια, το κλίμα. Για το κλίμα υποστηρίζουμε την ε, επενδύσεις σε πηγές ενέργειας ε, It's of course on reducing energy consumption χαμηλών εκπομπών. Η εξοικονόμηση ε, πόρων, η βελτίωση των ενεργειακών πηγών, η υποστήριξη των επιχειρήσεων, νέες πράσινες θέσεις η ευημερία των πολιτών είναι θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και οι επενδύσεις θα πρέπει να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση και με βάση την αρχή του ότι όλοι θα πρέπει να κερδίζουν από αυτό την σχέση. Αυτό φαντάζομαι ότι θα, πρέπει να είναι, θα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ωφελής για όλη την Ευρώπη. Όσον αφορά ε, αυτές τις επενδύσεις και τις επιπτώσεις επί των θέσεων απασχόλησης, βάσει μελετών υπολογίσαμε ότι κατά μέσον όρο η πολιτική συνοχή δημιουργεί 17.000 ε, θέσεις εργασίας, αν επενδυθεί ένα δις ευρώ και αν γίνουν και ενεργειακές επενδύσεις στα διάφορα κτίρια, θα δημιουργηθούν και πολλές άλλες θέσεις απασχόλησης. Οι επιπτώσεις λοιπόν είναι σαφείς Εάν λοιπόν οι επενδύσεις που γίνονται στα πλαίσια του, της πολιτικής συνοχής στοχεύουν στην ενεργειακή απόδοση και προστασία των κτηρίων, έχουμε και μία προστιθέμενη αξία. Κατά την άποψή μας, αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθεί στην πολιτική να μην υποχωρεί στο Συμβούλιο. Δεύτερο ε, θέμα, αφορά το ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιλέξουν ε, τον τομέα στον οποίο θα θέλουν να κάνουν επενδύσεις, να μην γίνονται όπως βλέπουμε μαζικές επενδύσεις στα δίκτυα δικών μεταφορών, όπου εδώ έχουμε να κάνουμε με μέσο μεταφοράς ε, το οποίο Τελευταίο θέμα που αφορά ε, την ε, ενέργεια και την προσοχή του περιβάλλοντος είναι τα ε, στερεά καύσιμα. Βλέπουμε ότι αντί να υποστηρίζονται νέες, νέοι ενεργειακοί πόροι και νέες ε, ε, πηγές ενέργειας πάλι υποστηρίζονται από το Συμβούλιο επιδοτήσεις για τα στερεά καύσιμα και πιστεύουν ότι το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να επιτρέψει κάτι τέτοιο. Στον κανονισμό IDF, πολύ σύντομα, πρέπει να πω ότι ασχολούμαι με τη βιοπικιλότητα και την αποδοτικότητα των πόρων που χρησιμοποιούνται η υποστήριξη των οικοσυστημάτων και των οικο... θα πρέπει να υποστηρίζονται. Τελευταίο στοιχείο έχει σχέση με τους δίκτες και στόχους που αφορούν το περιβάλλον Κάναμε κάποιες προτάσεις με κάποιους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς δείκτες που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο της ε, κανονισμού περιφερειακής πολιτικής, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τις απαραίτητες μετρήσεις και αν έχουμε τους κατάλληλους δείκτες, θα μπορούμε να δούμε και ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους θέλουμε να υλοποιήσουμε στα πλαίσια των επενδύσεων που γίνονται και στα πλαίσια της, των στόχων 2020. Τώρα, όσον αφορά τον κανονισμό της πολιτικής συνοχής, ένα θέμα αφορά την βιοπικιλότητα και την αποδοτικότητα των πόρων που χρησιμοποιούνται. Ζητείτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηριχθούν να υποστηριχθεί η πολιτική της Natura ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν όλες οι προτάσεις που αφορούν υλοποίηση της πολιτικής Natura 2000 και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να καταστεί σαφές στον κανονισμό. Τελευταίο στοιχείο, ο κανονισμός που αφορά το Ταμείο Συνοχής είναι προσανατολισμένος στους στόχους. Θα πρέπει να έχουμε έναν εμπεριστατωμένο κατάλογο των δικτών και των στόχων και των που θέλουμε να υλοποιήσουμε, να συμπεριλαμβάνουμε τους περιβαλλοντικούς στόχους όταν αυτό είναι δυνατόν, ώστε να γίνονται οι κατάλληλες επενδύσεις με τους δείκτες συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών δικτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Γκοντινό. Ο κύριος Πίτερ Μπέρκοβιτς από την Επιτροπή θέλει να λάβει το λόγο. Um, Σας ευχαριστώ. Να αναφερθώ και εγώ γενικότερα για το ρόλο που διαδραματίζουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσει τόσο για την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και για τι συζητήσει που γίνονται στου τριμερεί διαλόγου. Όπως ξέρετε, η γενικότερη ιδέα για τη μεταρρύθμιση της ε, πολιτικής συνοχής είναι ότι χρειαζόμαστε μια πιο αποτελεσματική πολιτική συνοχής, με καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερη διασύνδεση με τους στόχους Ευρώπη 2020 και ιδίως με τους επιμέρους στόχους στους οποίους αναφέρθηκαν οι ομιλητές. Έχουμε προτείνει λοιπόν νέους μηχανισμούς, είπαμε ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στις επιδόσεις, ότι θα πρέπει να θέσουμε συγκεκριμένες προϋποθέσεις στην αρχή της αιρεσιμότητας και είπαμε ότι χρειαζόμαστε όμως και πιο ισχυρές εταιρικέ σχέσεις. Για ποιο λόγο, καταρχάς, για τη χρηστή διακυβέρνηση, αλλά πέρα από αυτήν και για το ζήτημα της αποτελεσματικότητας, δηλαδή πώς τα διαθέσιμα κονδύλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και θα ήθελα να αναφερθώ και σε μια πρώτερη έκθεση που είχαμε, η οποία επέκρινε τη διαδικασία της Λισαβόνας, ακριβώς επειδή η διαδικασία αυτή δεν μπορούσε να συμπεριλάβει καλά στα διάφορα προγράμματα τους τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες. Υπάρχουν τώρα κάποια στοιχεία τα οποία ήδη έχουν αναφέρει οι προλαλήσαντε. Ενδεχομένω το πιο σημαντικό είναι ο κώδικα συμπεριφορά, Βέβαια τον κώδικα αυτό πρότεινε η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρούμε ότι είναι θεμελιώδου σημασία αν πραγματικά θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποια ελάχιστα πρότυπα και αν θέλουμε να προωθήσουμε τι βέλτιστε πρακτικέ. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι εξίσου σημαντικά, τα ανέφεραν αυτά και οι προλήσαντε. Καταρχά, community local development, να καταφέρουμε να έχουμε μία ανάπτυξη τοπικών κοινοτήτων. Αυτό προβλέπεται για όλα τα ταμεία και πιστεύω πραγματικά ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εμπλέξουμε περισσότερο τους τοπικούς φορείς προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Και βλέπουμε ότι στα πλαίσια του, ε, κοινωνικού, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης υπάρχει ακόμα ένα πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και εμπλοκής περισσότερων τοπικών φορέων. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κοινοτικά προγράμματα για να αντιμετωπίσουμε διάφορα κοινωνικά προβλήματα όπως η διακριτική μεταχείριση ή ο κοινωνικός αποκλεισμός. Όλες αυτές οι αρχές, όλοι αυτοί οι στόχοι δεν είναι θεωρητικοί, πρέπει να εφαρμοστούν και στην πράξη και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε ένα υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης, το οποίο βρίσκεται εκτός δημοσίου τομέα, αν θέλετε, βρίσκεται περισσότερο στα χέρια των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε τη γνώση των οργανώσεων αυτών. Υπάρχουν κάποιοι τομείς, τους οποίους αναφέρατε, όπου πραγματικά θεωρούμε ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις μπορούν να εκδραματίσουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση των προτεραιοτήτων μας και συμφωνώ με τα όσα είπατε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιους από τους τομείς αυτής. Ο πρώτος είναι ο τομέας της φτώχειας, της ένδυας και της κοινωνικής ένταξης. Προβλέπονται στα προγράμματα κάποιοι νέοι μηχανισμοί, δεν θα τους αναφέρω τώρα έναν προς έναν, Ουσιαστικά πάντως έχουμε πλέον ένα μηχανισμό για την καταπολέμηση της φτώχειας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό. Βέβαια έχουμε πολλούς διαθέσιμους πόρους για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κατοικιών. Πρέπει και οι πόροι αυτοί να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να επιτευχθούν οι στόχοι στους οποίους αναφέρθηκαν οι προαλήσαντες. υπάρχει και ένας νέος μηχανισμός που προτάθηκε κυρίως με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είχε κάνει και η Ευρωπαϊκή Επίτροπη μια αρχική πρόταση, αλλά επέμεινε ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το να εστιαστούμε περισσότερο στι δημοκρατικές, συγγνώμη, στις δημογραφικές αλλαγές να υπάρχει δηλαδή και δημογραφική διάσταση στα προγράμματα. Ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να αφαιρθώ σε ένα ακόμα τομέα που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και για τον οποίο εργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι συμφωνεί τελικά και το Συμβούλιο, το ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την όλη διαδικασία εμπλοκή των διαφόρων εταίρων πολύ περισσότερο στο μέλλον. Βλέπουμε ήδη στα πλαίσια των τριμερών διαλόγων ότι γίνεται μια όλο και μεγαλύτερη αναφορά στις εταιρικέ σχέσεις και γίνονται και πάρα πολλές αναφορές αξιολόγησης της συνεργασίας που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τους διαφόρους εταίρους της. Αυτό θα γίνεται πλέον σε αιτήσια βάση. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Ε, Σας ευχαριστούμε κύριε Μπερκόβιτς. Το λόγο τώρα έχουν συντονιστές από τις πολιτικές ομάδες. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Ο κύριος Βαν Νιστερόι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, ομιλητές για όλες αυτές τις παρεμβάσεις τους. Πιστεύω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε όλες αυτές τις πληροφορίες και τουλάχιστον όσες λάβαμε κατά τη διάρκεια του τελευταίου του ήταν πάρα πολύ σημαντικές και αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτηση στις διάφορες ομάδες εργασίας και καταφέραμε τελικά να διαμορφώσουμε ή θα διαμορφώσουμε καλύτερα την πολιτική συνοχή στα επόμενα επτά χρόνια. Μία γενική ερώτηση προς όλους τους ομιλητές. Είναι καταπληκτικό να έχουμε πολύ σύντομα μία συμφωνία για τους διάφορους αυτούς κανονισμούς. Αλλά εσείς τι πιστεύετε ότι συμβαίνει στα επιμέρους κράτη-μέλη τη στιγμή που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις πρώτες συμβάσεις, τις πρώτες συμφωνίες εταιρικέ σχέσεις, Βλέπουμε ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν ήδη το πρώτο σχέδιο, το δεύτερο σχέδιο της συμφωνίας αυτής διαθέσιμο. Στην πράξη όμως, τι γίνεται. Οι εταίροι σας, οι οργανισμοί που συμμετέχουν στις δικές σας τις ομοσπονδίες πραγματικά συμμετέχουν στην όλη αυτή διαδικασία, είναι ήδη έτοιμοι, γιατί το 2014 δεν είναι μακριά και θα πρέπει να προετοιμάσουμε τα προγράμματα με τον νέο αυτό τρόπο. Τι συμβαίνει λοιπόν επί τόπου, στις πόλεις, στις περιοχές, στις περιφέρειες, στις χώρες στις οποίες εκπροσωπείτε. Είστε σε επαφή με τις δημόσιες αρχές, πώς προχωράει η διαδικασία γιατί αν είστε ικανοποιημένοι με την ενεργειακή αποδοτικότητα, με τα προγράμματα στέγασης, με την διάσταση ε, τη δημογραφική, με την ε, ενεργογύρανση, ε, θεωρείτε ότι όντως όλα αυτά αποτελούν πραγματικότητα πλέον στα διάφορα κράτη-μέλη. Θα μπορέσουν πραγματικά τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν προγράμματα σε όλους αυτούς τους τομείς το επόμενο χρονικό διάστημα. Και έπειτα, η σχέση ανάμεσα στους νέους αυτούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως το είπα, ο μηχανισμός Πρωταξιακή βοήθειας ή τα προγράμματα για την ενεργογύρανση. Θεωρείτε ότι υπάρχει τελικά μία διασύνδεση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές αυτές προθέσεις, αυτούς τους στόχους και την λήψη αποφάσεων και την έγκριση πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο πώς λειτουργούν τα πράγματα στην πράξη. Αυτό θα ήθελα να μάθω. Και πραγματικά νομίζω ότι έχουμε κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Αν δείτε πόσα πράγματα έχουμε τροποποιήσει αυτή τη στιγμή μέσω τροπολογιών που έχουμε υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε κύριε Βανίστερο. Το λόγο έχει κυρία Κλέβα. Mm, I Ήθελα να καλωσορίσω αυτή τη συζήτηση είναι νομίζω εκπληκτικό το πώς το βλέπουμε όλοι ε, από διαφορετική πτυχή το, το ίδιο έγγραφο αυτό. Οι και όσα είναι γνωστές, ε, λαμβάνουμε τις συνεισφορές σας τακτικά, όχι μόνο για τον κοινό κανονισμό, αλλά για κάθε έκθεση που έχουμε εδώ πέρα. Και πριν ε, χαμογελούσαμε πράγματι για την πλατφόρμα για τους ηλικιωμένους ε, πράγματι είχαμε λάβει εκατοντάδες ε, προτάσεις όταν μιλούσαμε για την πολιτική συνοχής για την επόμενη περίοδο. Δεν έχω ερωτήσεις. Θα ήθελα να ε, καλωσορίσω αφενός την πλατφόρμα, την Age Platform, γιατί δραστηριοποιούμε και στην Επιτροπή Γυναικών και εκεί πέρα βλέπω κάποια πράγματα. Τώρα για την κοινωνική στέγαση, ναι, γράφω και μια γνωμοδότηση σε σχέση με τις γυναίκες και θέλω βέβαια και τη συνεργασία σας στο μέλλον. Και θα ήθελα να μου δώσετε και το, το PowerPoint σε ηλεκτρονική μορφή. Γιατί το φωτοαντίγραφο δεν φτάνει, γιατί είναι, είναι ασπρόμαυρο και δεν, δεν μπορούμε να καταλάβουμε όταν θα μπορούσατε να μας το στείλετε και θεωρώ πραγματικά πως ε, η κοινωνική στέγαση είναι θέμα τοπικών και περιφερειακών αρχών. Δεν φαντάζεστε πόσες προτάσεις για τροπολογίες είχαμε για την πρόταση επίσης ενεργειακής αποτελεσματικότητας πέρσι και απευθύνομαι στο ΒΒΕΦ. Ε, είναι θέμα τοπικών ε, και περιφερειακών αρχών. Εμείς ε, κάνουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Γι' αυτό ήθελα να πω κάποια λόγια, γιατί νομίζω πως τελικά όλοι στην ίδια βάρκα είμαστε, όπως λέμε. Γιατί περιγράψατε όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα συζητάμε εμείς στην Επιτροπή μας, συνεχώς. Ευχαριστώ, κύριο Σρέντερ από τους Πράσινους. Ε, ευχαριστώ πολύ. Τρία πράγματα θέλω να πω. Ήταν ενδιαφέρον, όπως είπε η κυρία Περέν, για ότι χρειαζόμαστε ορθή ε, διακυβέρνηση. Ναι, καλό αυτό, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για διαπραγμάτευση με συγκεκριμένα θέματα, για συγκεκριμένες λέξεις με στην ε, νομοθεσία. Και ολοκληρώθηκε αυτή η διαπραγμάτευση χτες με την συζήτηση και μόνο μικρές α, ε, α, ε, τεχνικές αλλαγές αναμένονται. Αλλά βεβαίως εκεί πέρα είναι η υψηλή πολιτική αντιπαράθεση για αυτά τα μικρά τεχνικά ζητήματα ή λέξεις και με μονομένες λέξεις. Και εκεί πέρα θα ήθελα να μην παραμείνετε τόσο γενικοί στις δηλώσεις σας, αλλά συγκεκριμένα να μας πείτε τι θέλετε για να υπάρξει σωστή διακυβέρνηση. Και ένα ερώτημα προς τον εκπρόσωπο του, κύριου του ΒΒΕΦ, τον κύριο Γκοντάου. απευθύνεται επιστολή στα κράτη-μέλη, αλλά από το τριμερή διάλογο φαίνεται πως δεν, δεν την έλαβαν ποτέ. Δεν μπορεί και να μην τη διάβασαν, ναι, ναι. Κάπου στο δρόμο χάθηκε μεταξύ γραφείου σας και κρατών μελών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επανέρχομαι σε αυτά τα δευτερεύοντα ζητήματα και μικρές τεχνικές αλλαγές σε ένα κείμενο, σε ένα τριμερή διάλογο και θεωρώ έχουμε μόνο κάποιες ώρες για να επιδοθεί εκεί που πρέπει αυτή η επιστολή. Δεν ξέρω αν έχετε λεφτά για να το στείλετε σήμερα με courier ε, στην ε, Κυπριακή μόνιμη αντιπροσωπεία. Ε, αλλιώς δεν θα φτάσει νομίζω εκεί που πρέπει η επιστολή. Και το τρίτον αφορά το ερώτημα διοξίδιο του άνθρακα και βελτίωση κτλ. Και μια οικονομία χαμηλών εκπομπών. Το θέμα δεν αφορά μόνο την ε, στέγαση ε, αλλά και άλλα παράγματα. Είναι δηλαδή κάπως ανοιχτό το εάν θα εκμεταλλευτούν τα κρατημέλη αυτό το οποίο λέτε. Δηλαδή να κάνουν τα σπίτια έτσι πιο φιλικά προς την ενέργεια. Οπότε είναι ζήτημα εθνικού επίπεδου και έτσι ερχόμαστε πάλι στο ζήτημα εταιρική σχέση και συνεργασία και θα ήθελα να μάθω πώς θεωρούν οι εταίροι, πώς ε, πριν την προγραμματική διαδικασία θα μπορέσουν να συμπεριληφθούν για να μπορέσουν να ασκήσουν κάποια επιρροή. Και για να μπορέσει να γίνει αυτή η συνεργασία ακριβώς για την προγραμματική περίοδο. Τι πρέπει να γίνει τώρα έτσι ώστε αυτοί οι εταίροι να μπορέσουν να συνεισφέρουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Σρέντερ. Κύριε Σόλπρη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πάντα μπορούμε να αναρωτηθούμε μήπως θα είναι πολύ αργά πλέον να έρθουν οι εταίροι μετά από τις συζητήσεις που γίνονται στην Επιτροπή για τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ξέρω όμως ότι και οι εταίροι και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι πολύ καλά ενημερωμένοι, δεδομένου ότι αυτό είναι από την αρχή. Δηλαδή, αυτό ήταν στην αρχή πρόταση και ξέρουμε ότι μας παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς από την αρχή και ξέρουν τι, πώς προχωρούν τα πράγματα μέχρι σήμερα. Η παρουσία τους δεν ε, είναι για μένα να επαναλάβουμε αυτά τα οποία δεν ξέρουμε, αλλά να πείσουμε αυτούς που διαπραγματεύονται στο τελευταίο στάδιο να πολεμήσουν για να κατορθώσουν αυτό που θέλουν. Και ως συνήθως είναι οι εταίροι μας προετοιμασμένοι πολύ καλύτερα από πολλούς από εμάς, δεδομένου ότι δεν χάνονται στις γενικότητες, αλλά ξέρουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και μπορώ να πω ότι όσον αφορά το ADF, e ότι όντως γενικώ έγινε μία προσπάθεια στις θεματικούς στόχους να εισαρθεί το στοιχείο της δημογραφία, στο δημογραφικό στοιχείο, στους θεματικούς στόχους. Έχει συμπεριληφθεί. Όχι. Καταρχάς είχαμε την ε, πρωτοβουλία στην Επιτροπή μας, στην αρχή, αλλά δεν έγινε αυτό. Είναι πολύ αργά για να εισαγάγουμε τώρα το θέμα αυτό του δημογραφικού στοιχείου, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν κατάλαβα πολύ καλά ποια είναι η πρώτη πρόταση που έγινε για τον, την, από την πλατφόρμα αυτή και πώς μπορεί να ενισχυθεί. Όσον αφορά το Παγκόσμιο Ταμείο τη Φύση, πολλές φορές είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και υπάρχουν στοιχεία τα οποία υποστηρίζει η Επιτροπή μας και η Επιτροπή Ενέργειας, κυρίως αυτό της ανεργιακής απόδοσης και δεν συμμερίζομαι αυτό που είπε η συνάδελφος. Το θέμα της στέγασης είναι μεγάλο πρόβλημα, όλο και πιο οξύ πρόβλημα και μεγαλύτερο στο Κοινοβούλιο. Είπα ότι το θέμα αυτό είναι θέμα επιλογής των κρατών μελών, αν θέλουν να επικεντρωθούν στο θέμα της. Στα κράτη-μέλη δεν είναι ανόητα. Ξέρουν ποιες επενδύσεις είναι σχετικά απλές, γρήγορες και αποδοτικές. Το θέμα της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια είναι μία δράση ε, που έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και ταχύτητα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθεί να κάνει και ο κύριος Μποστινάρου. Και όπως θέλετε θέλουμε να επιτύχουμε σε διάφορα επίπεδα, σε κατώτερα επίπεδα στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής κάποια ποσόστα. 16-22 αντιστοίχως. Αντιθέτως, χρησιμοποιείται το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας και απόδοσης στον τομέα των μεταφορών, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι το αντίθετο. Θα πρέπει στο επίπεδο της στέγασης, αρχίζοντας από τα δημόσια κτίρια, να αρχίσουμε με την ενεργειακή απόδοση. Και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το επιλύσουμε και κυρίως να δούμε αν ε, ε, να μας πριν να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και να ξέρουμε επίσης τι γίνεται με τις ε, κρατικές ενισχύσεις που να δοθεί ακόμη για την ενεργειακή απόδοση. Ως εισηγητής, εγώ, έχω μία θέση η οποία ίσως δεν είναι αυτή της ε, Επιτροπής ή του Παγκοσμίου ε, Ταμείου για τη φύση όσον αφορά το θέμα των εκπομπών. Ρίου, πιστεύω λοιπόν ότι για να καταλάβουν καλύτερα στους θεματικούς στόχους, κυρίως το άρθρο 5, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ενεργειακή απόδοση είναι πάρα πολύ σημαντική. Επίσης, τι εννοούμε με τη στέγαση. Δεν θέλουμε να δώσουμε ορισμό στον εφαρμοστικό νόμο θα εξηγηθούν όλα αυτά. Ε, η στέγαση, κοινωνική στέγαση. Εμείς δεν θα πρέπει αυτό το πράγμα να το συμπεριλάβουμε στον κανονισμό. Κάτι με το οποίο διαφωνώ με τους ομιλητές είναι οι δείκτες. Πιστεύω ότι οι δείκτες που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικοί για την αξιολόγηση της ε, πολιτικής που κάνουμε δεν θα πρέπει να υπάρχουν στον κανονισμό, αλλά στον εφαρμοστικό κανόνα. Στον... Ε- Εάν μέσα στο κύριο κορμό του κειμένου, στο νομοθετικό κείμενο, εισαγάγουμε ε, την έννοια των ε, δικτών, δεν θα έχουμε ε, τα κατάλληλα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε κάτι το απόλυτα σαφές, αλλά νομίζω ότι, επαναλαμβάνω εγώ συζητητής, θα προτείνω να μην υπάρχει μνήα των δικτών, διότι κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, αν μιλήσουμε ε, για δείκτες που είναι κάτι το τεχνικό θα πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε διαπραγμάτευση από εδώ και από εκεί. Δεν είναι η θέση λοιπόν αυτού του θέματος που αφορά τους δείκτες που είναι τεχνικό μέσα στο νομοθετικό κείμενο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Όλμπριχτ. Τρεις ε, ερωτήσεις ακόμα έχουμε από τρεις ομιλητές και συνέχεια θα ακούσουμε και τις απαντήσεις. Ο κύριος Μποστινάρου πρώτος. Σας ευχαριστώ πολύ. Μετά από τα τόσα σημαντικά πράγματα τα οποία ακούσαμε, τα οποία ανέφεραν ε, οι συναδελφοί μου, το μόνο το οποίο μπορώ εγώ να προσθέσω είναι το ότι θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της ε, διαδικασίας σύνταξης ε, του σχεδίου έκθεσης με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Βλέπουμε πάρα πολύ τη συμβολή του σήμερα στο περιεχόμενο της έκθεσης. και όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας για την στέγαση, η συμβολή σας ήταν καταπληκτική πραγματικά. Και βλέπουμε για μία ακόμη φορά ότι κάθε φορά που μιλάμε για φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές, για την μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, για πράσινες θέσεις εργασίας, οι άνθρωποι από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι σε θέση να παρέχουν πάρα πολύ καλές προτάσεις στα πλαίσια μιας έκθεσης και ενός κανονισμού. Σα ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και ξέρω ότι ε, εκπροσωπώ στι ευχαριστήσει μου αυτές και τι διάφορες κοινότητες και τι περιφέρειες. Θα ήθελα επίση να στείλω τώρα ένα μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Θα πρέπει η διάσταση της εξοικονόμησης ενέργειας για τη στέγαση να υπάρχει σε πάρα πολλές πολιτικές προκειμένου να καταφέρουμε να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, προκειμένου να έχουμε και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για το ζήτημα της εξοικονόμησης της ενεργειακής και της θέρμανσης. Κατά αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουμε πολύ καλύτερες συνθήκες για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξέρω πολύ καλά ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσει έχουν διαδραματίσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να πείσουμε το Συμβούλιο εκεί πέρα που υπάρχει ακόμα αντίσταση από τι χώρε αυτέ, οι οποίε. ακόμα δεν έχουν πιστεί. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική συνεργασία και σας ευχαριστώ πολύ γιατί παρήχατε επίσης διατάξεις για το Natura 2000. Οι τροποποιήσεις αυτές είχαν και τη δική σας την υποστήριξη. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε κύριε Μποστινάρο, κύριος Βλάσεκ έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω τα όσα υπόθηκαν ήδη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας και από προσωπικής ε, εμπειρία μπορώ να πω ότι η συνεργασία μας βασίζεται στις πολύ καλές επαφές που έχουμε. Δεν αναφέρομαι μόνο σε απλές διαπραγματεύσεις, αλλά πολλές φορές και στη συνεργασία που είχατε εσείς με Intergroup του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως για παράδειγμα με την Διακομματική Ομάδα για την Αστική Ανάπτυξη, σε σχέση με αυτά που είπε ο Λάμπερτ Βανίστερόι. Πού έχετε εντοπίσει εσείς προβλήματα, πού θεωρείτε ότι δεν υπάρχουν ε, καλές ανταποκρίσεις, σε ποιο επίπεδο, είναι σε τοπικό, περιφερειακό, σε εθνικό επίπεδο, Υπάρχει αδυναμία συνεργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πετύχουμε συνένεση σε κάθε επίπεδο. Εγώ από την προσωπική μου εμπειρία γνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε συνένεση για πάρα πολλές πολιτικές, περιβαλλοντικές, αστικές, αλλά σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, περιφερειακό και εθνικό. Πού έχετε εντοπίσει εσείς προβλήματα, μπορείτε να μου το πείτε. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, όσον αφορά τις μεταφορές, πιστεύω ότι πάρα πολλές χώρες πρέπει να επενδύσουν στις μεταφορές. Από οικολογική όμω πλευρά θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες προκειμένου οι μεταφορές αυτές να είναι οικολογικά βιώσιμες. Και αυτό ισχύει πάρα πολύ για τις αστικές μεταφορές. Πρέπει να γίνουν εδώ οι κατάλληλες επενδύσεις γιατί καταλαβαίνετε ότι το αστικό περιβάλλον αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα. Χρειαζόμαστε λοιπόν τέτοιες φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις στις αστικές μεταφορές. Μεταφορές πάρα πολύ σημαντικές για όλες τις πόλεις. Χρειαζόμαστε τις μεταφορές, αλλά αυτές θα πρέπει να είναι βιώσιμες και οικολογικές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Βλάσεκ. Ο κύριος Μαρίζ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ να κάνω και εγώ με τη σειρά μου κάποιες παρατηρήσεις για τα σημεία τα οποία ακούσαμε από τον κύριο Γκοντινό που εκπροσωπεί το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση. Όταν έλαβα την αρχική του πρόταση, μάλλον την αρχική πρόταση της Επιτροπής για το Γενικό Κανονισμό, δεν μου έκανε καμία εντύπωση το περιεχόμενο έβλεπα ότι ε, μολονότι υπήρχαν πάρα πολλές ασυνέπειες, στις οποίες αναφερθήκατε, υπήρχε αν μη τι άλλο μια γενικότερη συνειδητοποίηση των προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τις κλιματικές αλλαγές, ότι πρέπει να μετριαστούν τα προβλήματα αυτά και ότι θα πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε. Από την άλλη, όσον αφορά την βιοπικιλότητα, ως προς αυτό πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά κενά, πάρα πολλές αδυναμίες που προσπάθησε να βελτιώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει να σας πω ότι η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή και συγκεκριμένα οι συνάδελφοι που διαπραγματεύονται στους τριμερείς διαλόγους διαδραμάτισαν πλήρως το ρόλο τους. Το είπατε και εσείς όσον αφορά το άρθρο 8, δηλαδή τις οριζόντιες αρχές, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό, το οποίο κατάφερε να σωματώσει τον στόχο της βιοπικιλότητας και νομίζω ότι αυτό θεωρείται πλέον και εκτιμένο σήμερα. Εκεί όμως που υπάρχουν ακόμα κενά είναι οι θεματικοί στόχοι. Και αυτό λέει πολλά βέβαια, γιατί στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέγεται ξεκάθαρα ότι πρέπει να προωθήσουμε την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων, να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να προωθήσουμε την εξορθολογισμένη χρήση των πόρων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σταματάει εκεί και δεν αναφέρεται καθόλου στο ζήτημα της βιοπικιλότητας. Και καθότι είναι παρούσα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να τους επενθυμίσω ότι έχουμε μπει στο έκτο κύμα εξαφάνισης των ειδών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναλάβει δράση. Επομένως πρέπει πλέον σε συστηματική βάση να ενσωματώνεται την προστασία της βιοπικιλότητας στις διάφορες πολιτικές, όπως ακριβώς γίνεται με τις κλιματικές αλλαγές όπου προσπαθείτε μέσω διαφόρων πολιτικών να τις μετριάσετε και να προσαρμοστείτε σε αυτές. Ευχαριστώ. Έχετε λοιπόν πολλές ερωτήσεις. Έχετε τον λόγο. κύριε Κοντινού, ίσως. Πρώτος. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις, τα σχόλια. Θα απαντήσω σε δύο ζητήματα. Το ένα για την αρχή της συνεργασίας και το άλλο για το περιβάλλον και το κλίμα. Ευχαριστώ την κυρία Σρότερ για τα σχόλιά της, πως κάπου χάθηκε η επιστολή μας. Ε, την έχουμε στείλει σε όλους τους υπουργούς συνοχής και εξωτερικών ε, των κρατών μελών και βεβαίως όπως φαντάζεστε δεν μείναμε σε μια επιστολή Ήμασταν σε επαφή με πολλά κράτη-μέλη για πάνω από ένα χρόνο για τη στήριξη αυτή της αρχής της ε, συνεργασίας. Είχαμε συναντήσει σε πολλές ε, χώρες ε, και με πολλές αντιπροσωπείες στις Βρυξέλλες. Είχαμε και κάποιες απευθεία επαφές με Γερμανία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία, Ελληνία, Σλοβακία, Σλοβενία και θα ξεχνάω κι άλλες. Οπότε προωθούμε το ζήτημα αυτή της αρχής της συνεργασία και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στο επίπεδο των κρατών μελών κτλ. Αλλά όπως ξέρετε, πολλές ε, κυβερνήσεις είναι αντίθετες ε, ε, με τον υποχρεωτικό κώδικα συμπεριφοράς γιατί θέλουν τα χέρια τους ελεύθερα για το πώς θα εφαρμόσουν αυτή την αρχή. Και το συζητήσαμε αυτό με πολλά κράτη-μέλη κάποια στοιχεία που έλεγα δηλαδή. γιατί υποτίθεται πως είχαν θεσμικά ή συνταγματικά προβλήματα για να αποδεχθούν το ότι το ευρωπαϊκό επίπεδο θα είχε άποψη για το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η αρχή στο εθνικό επίπεδο. Και για να απαντήσω στο ερώτημα του κυρίου Βλάσακ, σύμφωνα με τους συναδέλφους μας που είναι επιτόπου, το βασικό πρόβλημα που έχουμε σήμερα είναι στο εθνικό επίπεδο. Βλέπουμε πολλά κράτη-μέλη όπου χτυπάν την πόρτα και δεν θέλουν να την ανοίξουν από μέσα για να μας εξηγήσουν το ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και ο σχεδιασμός ε, των μελλοντικών τέτοιων προγραμμάτων. Σε πολλές χώρες δεν έχουμε ιδέα για τη διαδικασία, για το χρονοδιάγραμμα, πότε η ΜΚΟ θα κληθούν σε ακρόαση, πότε θα στείλουμε τις προτάσεις μας. Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα, ειδικά στι ανατολικέ χώρε το να συζητήσουμε τις ε, συμφωνίε αυτές και τα επιχειρησιακά προγράμματα για την πολιτική συνοχή με τα κράτη-μέλη. Ενώ όλα τα κράτη-μέλη ξέρουμε πω ε, τα έχουν συζητήσει αυτά. Οπότε, προφανές, προφανές είναι πως ε, το σε συνθήκες ανταγωνισμού για να υπάρχουν υποχρεώσεις των ε, κρατών μελών να συμπεριλάβουν τους ενδιαφερομένους ακόμα δεν έχει επιτευχθεί. Οπότε ζητάμε έναν υποχρεωτικό κώδικα συμπεριφορά που θα έχει ίσου όρου ανταγωνισμού για όλα τα κράτη-μέλη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κενά και η κατάσταση δεν είναι σωστή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουμε δει κάποιες ε, ορθές πρακτικές ε, σε κάποια κράτη-μέλη. Και βεβαίως είχαμε και επαφές με προβουλευτές, με συγκεκριμένες προτάσεις με βάση την εμπειρία μας. Το άλλο ζήτημα Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για τις επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα που είπε και ο Σόλμπριχ. Ε, το συζητήσαμε αυτό. Είναι ένα ζήτημα ευαίσθητο το να επιδοτούμε ή όχι ε, ορυκτά καύσιμα πλέον ε, στην Ευρώπη. Υπήρχε μια συζήτηση στην Επιτροπή Ρέτζη για τη συμβαστική τροπολογία που έσπασε σε δύο μέρη και έφυγε το κομμάτι που αφορούσε την επιδότηση ορυκτών ε, καυσίμων. Οπότε η Επιτροπή ήταν κατά του να δοθούν τα λίγα χρήματα της, ε, περιφερειακή της περιφερειακής πολιτικής για τέτοιες επιδοτήσεις. Και η Ευρώπη έχει κάνει πολλές δηλώσεις και έχει κάνει πολλές δεσμεύσεις ε, στους G20, στον ΟΗΕ, στις διασκέψεις κλιματικής αλλαγής Οπότε ταυτόχρονα το να επιδοτεί ορυκτά καύσιμα στο εσωτερικό δεν ε, ενισχύει την αξιοπιστία της Ευρώπης. Το δεύτερο στοιχείο είναι πως ε, αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε πως μπορεί να υπάρχουν πολλές επενδύσεις που προγραμματίζονται σε αέριο για την επόμενη δεκαετία. Έτσι μπορεί να υπονομευθεί η μέγιστη ανάπτυξη των ΑΠΕ και αυτή είναι μια ανησυχία που έχουμε, όχι για το 2020, αλλά για το 2050. Γιατί ε, αυτή τη στιγμή έχουμε επενδύσει σε αυτές τις υποδομές, αυτές τις υποδομές θα χρησιμοποιούμε για να γίνει απόσβεση της επένδυσης. Οπότε χρησιμοποιούμε τις υποδομές που υπάρχουν και αν έχουμε υποδομή για αέριο Βεβαίω ε, δεν θα υπάρχει μετά δυνατότητα για ανανεώσιμε. Και αυτό είναι το ζήτημα για το 2030-2050. Ε, και πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Και... Δεν δημιουργούν πολλέ δουλειέ επίσης εδώ τη Ευρώπη ε, σε σχέση με και ειδικά ακόμη περισσότερο σε σχέση με ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Γιατί δημιουργούνται εκεί πέρα τοπικέ δουλειέ. Κατά την άποψή μα λοιπόν Υπάρχει... Ισχυρά... Υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα. Εξάλλου, μην ξεχνάμε πως μιλάμε κυρίως για την Πολωνία, για ένα δισεκατομμύριο τέτοιες επιδοτήσεις σε ορεικτά καύσιμα. Οπότε η Πολωνία έχει αυτή τη στιγμή μεγάλη οικονομική ανάπτυξη. Αν θέλει να επενδύσει ένα δισεκατομμύριο στο φυσικό αέριο, μπορεί να το κάνει μόνη της χωρίς την πολιτική συνοχή ε, και τις επιδοτήσεις. Γι' αυτό θεωρούμε πως οι επιδοτήσεις πολιτικής συνοχής στην ενέργεια μπορούν να πάνε στη ΑΠΕ και στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα για να υποφεληθεί κάθε χώρα και περιφέρεια στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Κοντινό. Η κυρία Παρό. Ευχαριστώ πολύ. Θα επικεντρωθώ σε κάποιες ερωτήσεις και όχι σε όλες ιδιαίτερα σε αυτές που αφορούσαν My intervention in the beginning, uh, knowing that we are already getting to the final. Προσπαθούμε στο κείμενο να συμπεριληφθούν όλες οι νέες προσεγγίσεις και οι θέσεις που θα θέλαμε να συμπεριληφθούν. Γι' αυτό επικεντρώθηκα στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να οργανωθεί το πρόγραμμα και να δοθεί υποστήριξη για την συμμετοχή των Εταίρων. Πράγμα το οποίο θα δώσει προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη, πράγμα το οποίο πρέπει να τονιστεί ακόμη περισσότερο. Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για την απόδοση και την καλύτερα αποτελέσματα για τους πολίτες της Ευρώπης. Γι' αυτό είναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα. Και όλες οι ε, όλα τα μέσα θα πρέπει να έχουν ως στόχο την βελτίωση καινοτόμων ε, λύσεων ε, ώστε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις προκλήσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι για να μπορέσουν σε αυτές οι λύσεις, οι θετικές να ισορρεθούν και να είναι περισσότερο καλύτερες, θα πρέπει να υπάρξει μία δομή σε επίπεδο ευρωπαϊκό ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν διασυνδέσεις, να μάθουμε από τις βέλτιστες πρακτικές, από τα λάθη που γίνονται και από τις λύσεις οι οποίες εφαρμοζόμενες κάπου έχουν οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα και όσον αφορά την απόδοση, τη και τα κέρδη, τα οικονομικά, την προστασία του περιβάλλοντος κτλ. Όσον αφορά το δημοκρατικό στοιχείο. Είχαμε πάρα πολύ καλά συμπεράσματα από το Συμβούλιο ΕΠΣΟ, το οποίο προώθησε αυτή την προσέγγιση. Όπως είπα προηγουμένως έχουμε την ομοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών που ζητά να εστιαστεί η πολιτική συνοχή στο να βοηθήσει τις τοπικές αρχές να ανταποκριθούν στα δημογραφικά προβλήματα και προκλήσεις και βεβαίως αυτό είναι κάτι μας διασυνδέει και με άλλες κοινωτικές πολιτικές. Την ε, πολιτική και εταιρική σχέση για θέματα ε, καινοτομιών, ε, την βούληση που έχουν εκφράσει τοπικές αρχές να συμμετάσχουν σε όλη αυτή την, ε, σε αυτό το νέο εγχείρημα. Στην ε, δημιουργία νέων ε, ερευνών που θα πρέπει να γίνουν ώστε να ληφθεί υπόψη και το θέμα της ηλικία και να μπορεί κανείς προχωρώντας ηλικιακά να είναι σε καλή υγεία, όλα αυτά σε συνέργεια με άλλα προγράμματα όπως αυτό των Smart Cities, Φερρυπίν και άλλες πρωτοβουλίες που θα μας επιτρέψουν να βελτιώσουμε και να προωθήσουμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες οι οποίες μπορούν να ληφθούν σε τοπικό και γενικότερο επίπεδο. Για μας το πιο δύσκολο επίπεδο Ε, είναι η δημιουργία εθνικών προγραμμάτων για να υποστηριχθούν όλες οι προσπάθειες που γίνονται ε, σε τοπικό επίπεδο για θέματα ηλικιακά. Πρέπει να πω ότι έχουμε πάρα πολύ καλή υποστήριξη από την ε, Φιλανδία και την Ιρλανδία Όσον αφορά τη Γαλλία, θα πάω τώρα στο Παρίσι, δεδομένου ότι γίνεται μία διάσκεψη για το θέμα αυτό. Υπάρχουν ε, λοιπόν προγράμματα εθνικής στρατηγικής. Στην Πολωνία και στην Πορτογαλία επίσης αναλαμβάνονται τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και θέλουμε όλα αυτά τα καλά παραδείγματα του τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει που παρουσιάζονται στις διάφορες χώρες της Ευρώπης να τα εκμελευτούμε ώστε να υπάρχει στα πλαίσια της πολιτικής συνογής μεταξύ τοπικού, περιφερειακού και εθνικού επίπεδου να υπάρχει καλύτερος συντονισμός για να βελτιωθούν τα πράγματα στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε κυρία Πάρεντ. Πέντε λεπτά έχουμε μόνο στη θέση μας για τους δύο εμπειρογνώμονες. Κύριε Ντιγιόλα, θα είμαι πολύ σύντομος. Όσον αφορά την εταιρική σχέση και την ερώτηση του κυρίου Βανίστερο, τι γίνεται επί τόπου. Κοιτάξτε, όντως τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή προσπαθούν να ετοιμάσουν το σχέδιο συμφωνίας εταιρικής σχέσης με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν οργανισμοί στέγασης που συμμετέχουν. Εμείς είμαστε παρόντες σε 19 κράτη-μέλη και παρόλα αυτά σε δύο μόνο περιπτώσεις η δική μας η Ομοσπονδία συζητά σε εθνικό επίπεδο με τις κυβερνήσεις για την προετοιμασία του σχεδίου συμφωνίας εταιρικής σχέσης. Δεν απορρέει βέβαια κάποιος, κάποια υποχρέωση αυτή τη στιγμή από τον καονισμό, αλλά χωρίς μια τέτοια υποχρέωση καταλαβαίνετε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για φορείς που εκπροσωπούν τον τομέα της στέγασης, της κοινωνικής στέγασης και το τομέα του περιβάλλοντος να συμμετέχουν. Ξέρετε ότι γενικότερα απευθύνονται σε εταίρους από το τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης ή πολλές φορές απευθύνονται απλώς στην τοπική αυτοδιοίκηση. Καλό αυτό, αλλά δεν φτάνει. Απαντάω επίση κατά αυτόν τον τρόπο και στην ερώτηση τη κυρία Σρέντερ. Το άρθρο 5 του σχεδίου καονισμού για τι κοινέ διατάξει, τουλάχιστον ο συμβασμό τη Προεδρία αυτή τη στιγμή δεν είναι ικανοποιητικό. Πρέπει λοιπόν εσεί να κάνετε κάτι, θα πρέπει να περασπιστείτε τη δική σα τη θέση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπω σα είπα, να συναυθούν αυτέ οι εταιρικέ σχέσει, Όσον αφορά τώρα το άρθρο αυτό το οποίο αναφέρεται στην ενεργοποίηση των τοπικών φορέων, πάλι εδώ πέρα αναφερόμαστε πάρα πολύ έντονα στο ρόλο των κρατών μελών, ότι τα κράτη-μέλη αυτά είναι τα οποία θα καθορίσουν τα κριτήρια για την επιλογή των στρατηγικών, τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα συστήσουν την Επιτροπή Επιλογής για τη Στρατηγική. Δεν μας αρκεί αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να ενσωματωθούν επισήμως και στο επίπεδο αυτό οι εταίροι και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναλάβει δράση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να απαιτήσει την εμπλοκή αυτών των φορέων. Τελευταία παρατήρηση όσον αφορά τους δείκτες και απαντώ έτσι στην ερώτηση του κυρίου Όλμπριχτ. Εμείς δεν υποστηρίζουμε την ιδέα των κοινών δικτών, να μπουν δηλαδή αυτοί στο διατακτικό του κειμένου. Θα προτιμούσαμε οι δείκτες να μπουν στις κατεξισοδότηση πράξης και να μην και να αποφύγουμε κατά αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο να έχουμε κακούς δείκτες στο κύριο τμήμα του κανονισμού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε και να υπολογίσουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο των επενδύσεων. Προτιμούμε λοιπόν οι δείκτες αυτοί να μπουν σε άλλη νομοθετική πράξη και οι δείκτες αυτές να καταρτιστούν από τους τοπικούς φορείς. Δεν θα θέλαμε να παγιωθούν κάποιοι δείκτες στο κύριο τμήμα του νομοθετικού κειμένου. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντιγιόλ. Ο κύριος Μπέρκοβιτς έχει το λόγο. Θα είμαι σύντομος. Να πω μόνο το εξής. Ελπίζουμε να έχουμε θετικό αποτέλεσμα τις επόμενες μέρες. Ανεξαρτήτως από αυτό. Το ζήτημα της εταιρική σχέσης είναι αυτή τη στιγμή στο κέντρο της ε, πολιτικής και αυτό οφείλεται στη δουλειά της Επιτροπής σας, ε, των ΜΚΟ και των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Και θα είναι, δεν θα είναι δυνατόν πλέον τα κράτη-μέλη να το αγνοήσουν. Και η Κομισιόν ε, θα παρακολουθεί αυτό το ζήτημα και στην διαδικασία προετοιμασίας ε, των συμβάσεων αυτών, αλλά βεβαίως και όταν η Κομισιόν θα φροντίσει να συμμορφώνονται με τον κανονισμό. Ευχαριστώ. I would like... Θα ήθελα Συγγνώμη, πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη. Είχα την παρουσίαση της δικής μου έκθεσης στην ΕΚΟΝ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους που εκπροσωπούν τις ε, ΜΚΟ ε, και για την συνεργασία σας, ε, γιατί νομίζω πως όλοι οι συνάδελφοι εκτιμούν πάρα πολύ τον ακτιβισμό σας, το ότι έρχεστε, χτυπάτε την πόρτα και εξηγείτε πράγματα, αν δεν το κάνατε... Ε, πιο πριν δεν είναι η συνάντηση αυτή στην οποία θα λυθούν τα προβλήματα. Εντάξει, είναι σημαντικές οι ακροάσει, αλλά δεν λύνονται εδώ πέρα τα προβλήματα, λύνονται, η δουλειά γίνεται όταν έρχεστε και μα τα λέτε εσείς και πρέπει να μας βοηθήσετε και σε εφαρμοστικέ ε, πράξεις, ε, όλα αυτά πρέπει να τα παρακολουθήσετε, καθώ είναι μια διαδικασία που μπορείτε να επηρεάσετε. Ε, supplementary or complementary και συμπληρωματικές ε, πράξεις και διατάξεις. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και ευτυχία στο νέο έτος ε, και τώρα θα ήθελα να προσκαλέσω τους ε, συναδέλφους να προετοιμαστούν για την ψηφοφορία. Τώρα θα περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία και θα ήθελα εδώ μια καρέκλα δίπλα μου άδεια γιατί χρειάζομαι να βοηθώ εδώ δίπλα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 Πέρας. Okay, so we start... Μάλιστα, ξεκινάμε με την έκθεση Βλάσακ. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή, τροπολογία 4 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 5 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, τροπολογία 6 υπέρ, κατά. Να επαληθεύσουμε την 6, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, δεκτή. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 8 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 11 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Να επαληθεύσουμε την 11 μάλιστα. So, which you want to check? Sorry, I'm confused. I voted 11. Μα συγχωρείτε, την 11, την 11 ψηφίσαμε και νόμιζα ότι είχε περάσει. 11, 11. Α, επαληθεύουμε την 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Close? Yeah, close. Yeah, full. And it's largely rejected. Απορρίπτεται με διαφορά. 12 λοιπόν υπέρ κατά αποχές. Να επαληθεύσουμε τη 12. Δεκτή. Τροπολογία 13 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ, κατά αποχές 15 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 16 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Απορρίφθηκε, ναι. 18 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 19 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε 19 ναι δεκτή τροπολογία 20 υπέρ κατά παληθεύουμε την 20 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. 16 με 18 απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ. Α, προφορική τροπολογία μα. Είναι κάποιος κατά. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν την 23 όπως τροποποιήθηκε. Υπέρ. Κατά. Αποχές Δεκτή. 24 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 25 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. 31 in favor. υπέρ, 2 κατά γίνεται δεκτή. Οπότε περνάμε στην έκθεση του μας έτσι για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Υπάρχει λοιπόν μια συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προφορική τροπολογία. είναι κανείς κατά. Καταπίπτει. Τροπολογία 11 όπως τροποποιήθηκε υπέρ κατά αποχές δεκτή. Και τώρα λέτε πως δεν υπάρχει χωριστή ψηφοφορία. Τροπολογία 12 Μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τροπολογία 13 προφορική τροπολογία. Είναι κανείς κατά. Ποιο είναι υπέρ της κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 19 με προφορική τροπολογία είναι κανείς κατά. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 21 χωρι... χωριστή. Μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ κατά. Επαληθεύουμε το μέρος δεύτερο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 18 με 18. Έτσι έχει απορριφθεί το μέρος δεύτερο. Συμβαστική 4. Όχι. Επί της διαδικασίας. Είστε υπέρ. Άρα εγκρίνεται. να επαναλάβουμε την ψηφοφορία για το δεύτερο μέρος της ε, τροπολογίας 21. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Εντάξει τώρα. Πέρας. Πάλι το ίδιο αποτέλεσμα, 18-18, ισοψηφία απορρίπτεται. Κάποιος άλλαξε, μετέβαλε άποψη. Απορρίπτεται, ναι. Μα το είδα, το είδα, ήταν ψήφισε, είδα το πράσινο λαμπάκι, εγώ το είδα. Όχι, με, με συγχωρείτε. Μα συνάδελφοι, ε, βλέπω. Ήταν ένα πράσινο λαμπάκι, ε, η συνάδελφος ψήφισε. Δεν ξέρω τι αφορά αυτή η τροπολογία, αλλά δεν, δεν πέρασε. Λοιπόν, συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 22 υπέρ, 24 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. πέρας. 33 με 3 συγχαρητήρια. Περνάμε τώρα. Λοιπόν, Μόησα Κλέβα, Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Συντονισμού των Οικονομικών Πολιτικών. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4. Χωριστή ψηφοφορία. Ποιο είναι υπέρ του πρώτου μέρου, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, ηλεκτρονική επαλήθευση, αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 με προφορική τροπολογία. Είναι κανείς αντίθετος. Όχι, το ψηφίζουμε ως έχει. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 η ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται με 17 προς 19. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20. Προφορική τροπολογία. Είναι κανείς αντίθετος. Όχι. Την ψηφίζουμε. Έτσι όπως έχει τροποποιηθεί. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 23 χωριστή ψηφοφορία, πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο μέρος υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση του δευτέρου μέτρου στις 23, αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται με 16 προς 22. Τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26. Προφορική τροπολογία. Είναι κανείς αντίθετος. Εάν όχι ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση της 26. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Όχι, απορρίπτεται με 14 προς 22, διορθώνει η Πρόεδρος. Απορρίπτεται. Ευτυχώς πεπαγρυμπρίνης Λαουμπέρ. Τρο... Ε, συμβιβαστική έξι Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία του σχεδίου γνωμοδότησης. Ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει ψηφοφορία, λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 35 προς 2. Εγκρίνεται λοιπόν. Και τώρα Περνούμε στην έκθεση τη κυρία Κόλαρσκα Μπομπίνσκα. Ο ρόλο πολιτική συνοχή Ευρωπαϊκή Ένωση και των φορέων τη όσον αφορά την εφαρμογή τη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική. Είστε έτοιμοι. Τροπολογία 1. Τη σύτρε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, υπόδειξη 5 της Ήτρε. Υπέρ κατά αποχές ε, ε, 34, καταπίπτει παραγραφός 2, 34 λοιπόν τροπολογία, υπέρ κατά, ας κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση, αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται με 26 προς 14. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παρά, ε, τροπολογία 43 υπέρ κατά. Νομίζω ότι απορρίπτει αλλά θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Λαμπέρ, για σένα τα κάνω όλα αυτά. Λίγη ψηφοφορία. 23 προς 12. Εγκρίνεται. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση Συμβιβαστικής 4. Αρχίζει η ψηφοφορία. 21 προς 18 εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Υπόδειξη 3 της Ήτρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 55. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται με 14 προς 26. 53. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση της 53. Λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται με 20 προς 18. Υπόδειξη 6 της Ήτρε. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 της Ήτρε. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο μέρος. Υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση του πρώτου μέρους. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 25 προς 13 εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Υπόδειξη 7 της Ήτρε. Γιατί λέγονται suggestions, υποδείξεις, υποδείξεις κάνουν μόνο. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62. Υπέρ, κατά, η ηλεκτρονική επαλήθευση της 62. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Με 25 προς 12. 63. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική. Όχι. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ε, συγγνώμη, το δεύτερο μέρος της συμβαστικής 7 δεν ψηφίσαμε. Ο Μιγγέλ θέλει ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 26 προς 14. Λοιπόν, και πάλι γυρίζουμε στις τροπολογίες. 69 υπέρ, κατά, ηλεκτρονική επαλήθευση. 27 προς 13 εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 88. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά νομίζω ότι εγκρίνεται. Ας κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν της 98. Λίγη ψηφοφορία και εγκρίνεται με 21 προς 16. 96. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση 96. Αρχίζει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 25 προς 11. 99. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση 102. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 19 προς 18. 104. Υπέρ. Σοσιαλιστές είστε υπέρ, εντάξει, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12, χωριστή ψηφοφορία, το πρώτο μέρος, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 111, υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση, αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική δεκατεία. Προφορική τροπολογία. Είναι κανείς κατά. Όχι. Την ψηφίζουμε έτσι ως έχει. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκατόν δεκαεπτά. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση 117. Λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται. 118. Υπέρ, κατά. Νομίζω ότι είναι η ίδια πλειοψηφία, πλειοψηφία αλλά ας κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθηση. 118. Λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται. 119. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 120. Υπέρ, κατά ηλεκτρονική επαλήθευση 120. Εγκρίνεται. 121. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση της 121. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται με 18 προς 21. 122 υπέρ κατά αποχέα συγκρίνεται, 123 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση 123 αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται με 18 προς 21. 124 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 126 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 13 ε, της ίτρα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 127. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία της 128. Αν δεν υπάρχουν ε, αντίθετα, ψηφίζουμε με χωριστή ψηφοφορία το πρώτο μέρος. Εγκρίνεται το δεύτερο μέρος. Εγκρίνεται. 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 132 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση υπέρ Α, συγγνώμη, αρχίζει η ψηφοφορία, λίγη η ψηφοφορία, εγκρίνεται. Εκατόν τριάντα τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται νομίζω. Λοιπόν, ε, κριτικό 3. Τροπολογία 2. Σε τελειωτικές σκέψεις. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ, κατά, Νομίζω ότι απορρίπτεται. Ναι, ναι, θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Για την 10 αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές Οι φιλελεύθεροι και οι σοσιαλιστές κατά του ECR και του ΕΛΚ, ποτέ κανείς δεν ξέρει Πώ θα εξελιχθεί το αποτέλεσμα τη πληροφορία. Λοιπόν, η ηλεκτρονική επαλήθευση 15. Για να δούμε, για να δούμε τι θα δούμε. 18 προς 18. Γι' αυτό ποτέ δεν καταλαβαίνω, λέει η πρόεδρος. Δεν ψήφισε κάποιος. Α, αυτός που δεν ψήφισε λοιπόν είναι υπέρ. Λοιπόν, για να ξαναεπαναλάβουμε, διότι αρχίζει η ψηφοφορία. Στην τροπολογία 15. Ψηφίσατε όλοι, έληξε ψηφοφορία. 19 προς 19! Άντε, πάλι απορρίπτεται. Πρέπει να εξασκηθείτε πριν από την ψηφοφορία. Τέλο πάντων, 16 υπέρ, κατά. Πάλι πολύ κοντά τα αποτελέσματα υπέρ και κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση υπέρ. Ε, συγγνώμη, αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υποδείξεις τη Ήτρε. Και τροπολογία 2. Τροπολογία 2, δεύτερο μέρος, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 4 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 9 καταπίπτει. 10 καταπίπτει. Καταπίπτει και η 11 και η 14. Λοιπόν, Υπόδειξη 15 της Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τελική ψήφος, ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 22 προς 17. Ολοκληρώσαμε την ε, ώρα της ψηφοφορίας. Κυρία Κολάσκα Μπαμπίνσκα, θέλετε να πείτε κάτι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιάδες που συνεργάστηκαν μαζί μου για τις συμβαστικέ τροπολογίες, όλους όσους μας έδωσαν πολύτιμες συμβουλές, ο κύριο, τον κύριο Βανίστελ Ρόι που με βοήθησε και όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μου. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν. Συνάδελφοι, αρχίζουμε τώρα πολύ σημαντικές ε, εκθέσεις από τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Όσοι λοιπόν θέλουν να ακούσουν τι έχουν να πούν, ας παραμείνουν στην αίθουσα και να σταματήσουν οι επιμέρους συζητήσεις. Lambert, you are reporting now. Lambert, έχεις το λόγο. Θέλω να σου το λόγο, αλλά δεν μπορώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε τώρα με τις κοινέ διατάξεις. Δεν έχω να πω τίποτα. Θα σας ενημερώσουν οι υπεύθυνοι συναδελφοί μας για το ποιοι τριμερείς διάλογοι έχουν λάβει χώρα, τι έχει συμβεί. Πρώτος ο Λαμπέρ, λοιπόν, Βανίστερόι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προσπαθώ να βάλω τα πράγματα σε μία σειρά. Ξέρετε ότι στην πολιτική υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές οπτικές γωνίες για διάφορους τομείς ε, όπως ε, η ενέργεια. Και εν γέννη πιστεύω ότι στην Ολομέλεια έχουμε και τον απαραίτητο χρόνο πλέον για να συζητήσουμε τέσσερις από τις εκθέσεις μας. Ορισμένε έχουν μόλις μάλλον εγκριθεί. Είναι πολύ καλό λοιπόν το ότι έχουμε συζήτηση, ότι προβλέπεται συζήτηση στην Ολομέλεια. Λοιπόν, επανέρχομαι τώρα στην νομοθετική εργασία για τους κανονισμούς μας. Να σας πω καταρχάς ότι χθες είχαμε την τελική ανταλλαγή απόψεων με τον αρμόδιο υπουργό της Ελλάδος, λέει ο πρόεδρος, της Κύπρου διορθώνει, Ήμασταν πολύ διαλλακτικοί και φιλικοί μαζί του, τον ευχαριστήσαμε για τη συμβολή του. Ήταν ειλικρινής βέβαια στάση μας αυτή, αλλά βασικά εκπροσωπούσε τη θέση του Συμβουλίου. Και ξέρετε ότι με το Συμβούλιο χρειάστηκε να κάνουμε πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις προκειμένου να τους φέρουμε στη δική μας την θέση. Η όλη διαδικασία δεν ήταν εύκολη. Πρέπει να σας πω ότι δέκα τριμερείς διάλογοι έλαβαν χώρα και αν είχαμε και τον 11ο σήμερα το βράδυ, ουσιαστικά καταλαβαίνετε ότι η διαδικασία δεν είναι καθόλου εύκολη. Είναι πολύ θετικό πάντως ότι στην εντολή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ενωμένο στην προσέγγιση. Ήταν πάρα πολύ καλό ότι καταφέραμε να είχαμε την ψηφοφορία αυτή τον Ιούλιο και ότι είχαμε ιδιαίτερα ισχυρή υποστήριξη. υποστήριξη με συγχωρείτε, δεν υπήρξε καμία εσωτερική διαμάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχαμε λοιπόν την εντολή αυτή στα χέρια μας και ξέραμε ότι θέλαμε να έρθουμε εδώ με θετικά αποτελέσματα στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Και ελπίζουμε ότι στην πρώτη συνεδρίαση που θα έχουμε τον Ιανουάριο με το νέο έτος θα έχουμε πλέον εγγράφος όλα αυτά τα αποτελέσματα, ένα τελικό κείμενο στα χέρια μας. Σήμερα αυτό το οποίο θα κάνω είναι να σας κάνω μία γρήγορη ανασκόπηση των σημείων στα οποία έχουμε καταλήξει στις διαπραγματεύσει και σήμερα στις, το βράδυ θα έχουμε ένα ακόμα τριμερή διάλογο που θα έχουμε μία μερική συμφωνία για τα σημεία εκείνα δηλαδή τα οποία έχουμε επεξεργαστεί στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού. Κωνσταντσε, θα αναφερθώ σε κάποια σημεία και όταν κουραστώ θα σου δώσω το λόγο να διαπραγματευτούμε και επ' αυτού κάποια στιγμή. Συνειδητοποιεί κανεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργάζεται με άλλους συναδέλφους. Στην διαπραγματευτική ομάδα ήμασταν εμείς οι δύο. Είχαμε βέβαια και την υποστήριξη της Προέδρου μας, της κυρίας Χούμπνερ, την ε, βοήθεια των σκιωδών εισηγητών και του προσωπικού μας που μέρα βράδυ εργαζόταν για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Εργαστήκαμε πάντως όλοι πάρα πολύ και εκτός ωραρίου αν θέλετε. Πώς έχουν λοιπόν αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Πρώτον, Ποιος είναι ο τίτλος που θα χρησιμοποιήσουμε, ποια είναι η ονομασία που θα δώσουμε στα ταμεία μας τα επόμενα 7 χρόνια. Αν δείτε τον ε, γενικό κανονισμό, βλέπετε ότι δεν υπάρχει κάποια νέα ιδέα ουσιαστικά. Βέβαια, τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι στιγμή δεν είναι θετικά για του Ευρωπαίου πολίτε και του εταίρου μα. Πιστεύω λοιπόν ότι σήμερα το βράδυ θα καταφέρουμε να καταλήξουμε στην ονομασία που πρότεινα εγώ και η Κωνσταντσε εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενδεχομένως να μιλήσουμε για ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Περιμένω ότι θα γίνει αποδεκτή η πρόταση αυτή. Ξέρετε ότι τα διαρθρωτικά ταμεία συνδυάζονται, σχετίζονται με τη συνοχή, αλλά αυτό που είπαμε και πάρα πολλές φορές και στην Ολομέλεια και στις συζητήσεις που κάνουμε εδώ πέρα στην Επιτροπή μας και σε πάρα πολλά εγγραφά μας, είναι το ακόλουθο, ότι ακολουθούμε μία πολιτική επενδυτική. Επομένως, Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Επενδυτικά Ταμεία, η ονομασία αυτή θεωρούμε ότι μας καλύπτει. Έχουμε ένα γενικό κανονισμό για τα πέντε ταμεία και ενδεχομένω να καταφέρουμε να εγκρίνουμε αυτή την ονομασία. Αυτή είναι αν μη τι άλλο η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έπρεπε να διευκρινίσουμε και πολλά πράγματα στο άρθρο 2, όσον αφορά τους ορισμούς δηλαδή. Και προσπαθήσαμε να προωθήσουμε και τη δική μας συνοπτική γωνία όσον αφορά την μακροπεριφερειακή στρατηγική. Και να πούμε ότι υπάρχουν και κάποιες συστάσεις προς συγκεκριμένες χώρες, κάποιες συστάσεις που λαμβάνουν υπόψη τον ιδιάζοντα χαρακτήρα ορισμένων κρατών μελών. Θεωρούμε λοιπόν ότι στο πρώτο έγγραφο έχουμε μια καλή ισορροπία. Δηλαδή, αναφερόμαστε στα εθνικά προγράμματα των κρατών μελών και έχουμε και ειδικέ συστάσεις προς τα κράτη-μέλη, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές. Το άρθρο 4 στη συνέχεια αναφερόμαστε εδώ στην ε, συμφωνία εταιρικής σχέσης και στις αρχές που θα πρέπει να διέπουν αυτές οι συμφωνίες. Υπάρχει εδώ πέρα μια γενική προσέγγιση η οικονομική, κοινωνική, εδαφική συνοχή, μια ολοκληρωμένη δηλαδή προσέγγιση. Και ουσιαστικά αυτό που λέμε προς τους εταίρους μας, αυτό που λέει ουσιαστικά το Συμβούλιο, δική του πρόταση είναι, μην επιφέρεται περισσότερο διοικητικό άχθος για όλους τους δικαιούχους των προγραμμάτων αυτών και όλους τους φορείς που καταρτίζουν αυτά τα προγράμματα. Μία σημαντική εξέλιξη έχουμε στο άρθρο 5. Χίλιες φορές θα μπορούσα να το πω αυτό εδώ στην Επιτροπή μας. Δεν θα έπρεπε να καταλήξουμε σε μία επανεθνικοποίηση της πολιτικής, της περιφερειακής πολιτικής. Τα ταμεία τα οποία μας απασχολούν είναι ειδικά ταμεία, στοχευμένα ταμεία, τα οποία έχουν να κάνουν με την περιφερειακή πολιτική. Εκεί απευθύνονται. Καταλήξαμε λοιπόν εμείς σε μια πολύ σκληρή προσέγγιση. Θέλαμε να έχουμε ένα ειδικευμένο έγγραφο όπου να αντικατοπτρίζεται και η τοπική αυτοδιοίκηση, η εκλεγμένη δηλαδή σε τοπικό αστικό επίπεδο. Το πετύχαμε αυτό. Έπρεπε βέβαια να διαπραγματευτούμε και με το Συμβούλιο. Δεν καταφέραμε να το περάσουμε αυτό σε σχέση με το Συμβούλιο. Πετύχαμε όμως έναν ορισμό όσον αφορά τις συμφωνίες, συμβάσεις, εταιρική σχέσεις. Είναι το βασικό έγγραφο το οποίο θα ισχύει τα επόμενα 7 χρόνια. Και στο έγγραφο αυτό έχουμε την τοποθέτηση των πόλεων, των περιφερειών, κυρίως της τοπικής αυτοδιοίκηση και έχει συμπεριληφθεί η συμβολή του στο έγγραφο αυτό. Δεν πρόκειται για ένα ξεχωριστό έγγραφο, πρόκειται για το πρώτο επίσημο έγγραφο το οποίο θα διέπει την εταιρική σχέση, αυτές οι συμφωνίες εταιρική σχέσης. Πετύχαμε εκεί πέρα ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να πετύχουμε και στη συνέχεια καταφέραμε να πετύχουμε και μία διατύπωση που ήθελε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να καταφέρουμε να εμπλέξουμε και άλλους φορείς. Υπάρχουν πάντως δύο επίπεδα αυτή τη στιγμή στην προσέγγιση. Αυτό ακριβώς θέλαμε από την αρχή. Και είναι πολύ σημαντικό να ισχύσει αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε και κατά την προεκλογική περίοδο για τις ευρωπαϊκές εκλογές δηλαδή, ότι απευθυνόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλο και περισσότερο σε μία αποκεντρωμένη διαχείριση. Εμπλέκεται όλο και περισσότερο η τοπική αυτοδιοίκηση. Το Συμβούλιο στη συνέχεια δεν ήθελε να διαγράψει τίποτα από τις διατάξεις που έχουν να κάνουν με την κατάρτιση των ε, συμφωνιών εταιρική σχέση, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέμεινε πάρα πολύ στο ζήτημα του κώδικα συμπεριφορά. Είπαμε ότι ο κώδικα αυτό θα πρέπει να αποτελεί ένα νομικό κείμενο το οποίο να ενσωματώνεται στον κανονισμό. Και θέλαμε λοιπόν το, το Συμβούλιο να αποδεχθεί τον κώδικα διοντολογίας, τον κώδικα συμπεριφοράς. Χαρήκαμε πάρα πολύ όταν είδαμε ως διαπραγματευτές ότι τελικά το Συμβούλιο συμφώνησε με την προσέγγιση αυτή. Συνέβαλε πάρα πολύ και η Επιτροπή των Περιφερειών ως προς αυτό. Καταφέραμε λοιπόν να το περάσουμε αυτό και υπάρχουν κάποια εκκρεμή ζητήματα ακόμα, θα τα διευθετήσουμε σήμερα το βράδυ. Ξέρετε πάντως ότι ήμασταν πάρα πολύ ισχυροί προσπαθώντας να προωθήσουμε τον κώδικα συμπεριφοράς, τον οποίο τελικά αποδέχτηκε το Συμβούλιο. Και είπαμε λοιπόν στο Συμβούλιο, κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή ήδη προετοιμάζουμε την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης. Το Συμβούλιο μας λέει ότι αν την προετοιμάσουμε τώρα τη συμφωνία αυτή, και αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τελικά τον Ιούλιο τους κανονισμούς αυτούς, ενδεχομένως και νωρίτερα, πιστεύω πάντως ότι όλοι αυτοί οι κανονισμοί μέχρι να γίνουν και οι μεταφράσεις και το καθεξής, μάλλον θα εγκριθούν τελικά τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε πάρα πολλές χώρες θα έχουν ήδη προτιμάσει τα έγγραφα εταιρική σχέσης. Θα βρίσκονται στο πρώτο σχέδιο, στο δεύτερο σχέδιο Επομένως τα κράτη αυτά μας λένε δεν θα πρέπει εμείς να τιμωρηθούμε στη συνέχεια αν τελικά δεν καταφέρουμε να συμπεριλάβουμε συμφωνίες αυτές όλες τις λεπτομέρειες που ενδεχομένω να εγκρίνει αργότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Απευθύνθηκα λοιπόν σε εμά και τους είπαμε εμείς ότι όντως μπορούμε σε ένα πρόσθετο έγγραφο με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά από πρόθεση με πρόταση με συγχωρείτε του Συμβουλίου να έχουμε ένα έγγραφο στο οποίο θα λέγεται ότι δεν θα χρειάζεται τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν από την αρχή της διαπραγματεύση για τη Συμφωνία εταιρικής σχέσης, αν τυχόν στο πρώτο ή στο δεύτερο σχεδιό τους δεν έχουν συμπεριλάβει όλα τα στοιχεία τα οποία θέλουμε εμείς. Μια τελευταία παρατήρηση να κάνω. Κουράστηκα και λίγο, το καταλαβαίνετε αυτό. Ε? αποδεχτήκαμε να ονομάζονται αυτές οι εταιρικέ σχέσεις contract agreement, συμφωνία σύμβασης. Το Συμβούλιο το αποδέχτηκε αυτό. Ουδέποτε είχε γίνει βέβαια κάτι τέτοιο με κανέναν, ούτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε θεσμικά όργανα, μα είπε το Συμβούλιο. Δεν μπορούμε να μιλάμε αυτή τη στιγμή για σύμβαση, για συμφωνία σύμβαση. Θα έχουμε λοιπόν στο μέλλον μια συμφωνία εταιρική σχέση, συμφωνία εταιρική σχέση που θα έχει όμω το περιεχόμενο το οποίο σα περιέγραψα. Κωνσταντσε, μπορεί να δώσει περισσότερε λεπτομέρειε γι' αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι, ότι κουράστηκε, Λάμπερτ, αλλά ευχαρίστω να λάβω εγώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις πριν ε, περάσουμε στα συγκεκριμένα. Χτες ήταν ε, η στιγμή της ευγένεια. Σήμερα νομίζω πως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Οι διαπραγματεύσεις με την πρόεδρη ήταν πολύ δύσκολες και κατά την άποψή μας αυτό οφείλεται στο ότι δεν σκέφτηκαν ποτέ τα κρατημέλη ότι έπρεπε να διαπραγματευτούν με το κοινοβούλιο. Δεν τους είχε περάσει από το μυαλό ότι θα μπορούσαν να απομακρυνθούν λίγο από την έντολή τους. Πέρασε καιρός μέχρι να μπει στο μυαλό τους ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Ε, και όταν λέει συμβιβασμό το Συμβουλίο εννοεί κάτι διαφορετικό από μας. Δηλαδή αυτοί εννοούν ε, τι μπορούμε, εμείς λέμε τι μπορούμε να πάρουμε να δώσουμε και ισορροπημένα. Για το Συμβούλιο συμβιβασμός είναι το Κοινοβούλιο να δεχτεί αυτά τα οποία αποφάσισε το Συμβούλιο. Και χρειάστηκε χρόνος για να έχουμε πραγματικές διαπραγματεύσεις. Και είχε προσπαθήσει και η Προεδρία να συνομιλήσει με μεμονωμένα άτομα. Δεν τα δεχτήκαμε αυτά. Γιατί βεβαίω θα έχει δυνατήσει πάρα πολύ και εξασθενήσει η θέση του Κοινοβουλίου και το επαναλαμβάνω. Θεωρώ πως με τη συμφωνία που επιτύχαμε για το στρατηγικό προγραμματισμό έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο και δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με τις διαπραγματεύσεις ε, του τριμερούς διαλόγου για τους συγκεκριμένους κανονισμούς. Είναι δύσκολες αλλά είναι πολύ πιο πολύπλοκος ο γενικός κανονισμός και περιέχει πάρα πολλά σημεία τα οποία δεν θέλει πολιτικά το Συμβούλιο. Και ακριβώς ε, γι' αυτό ε, είναι το δύσκολο το να θέλει να περάσει κάτι το Κοινοβούλιο. Τώρα ο Λάμπερτ αναφέρθηκε ήδη στον ε, κώδικα συμπεριφοράς. Τώρα μπορώ να επεκταθώ στο άρθρο 14 και 15 εγκρίθηκε το περιεχόμενο του κώδικα συμπεριφοράς, είναι μια πράξη κάτω εξουσιοδότηση και εδώ πέρα ε, αναμένω το τι θα γίνει απόψε έχουμε έξι ή εφτά διαφορετικές προτάσεις από πλευράς Συμβουλίου. Θεωρώ πως το Κοινοβούλιο νομίζω είχε, την, ε, είχε μια συμφωνία για την πρόταση παριθμών 5 για το καθεστώς και την προηγούμενη εβδομάδα, Τετάρτη, 9 η ώρα το βράδυ νομίζω έγινε αυτό. Εάν λοιπόν Ε, αλλάξει ξανά θα υπάρξει πραγματικά πρόβλημα. Δηλαδή, εάν πραγματικά καταστεί κενό γράμμα ο κώδικας συμπεριφοράς θα ε, είναι κάτι το απαράδεκτο και δεν το θέλει αυτό το κοινοβούλιο. Και εμείς είχαμε συμφωνήσει να υπάρξει διαχωρισμός στην εταιρική αυτή συμφωνία μόνο εάν δεχτεί ο το Συμβούλιο ένα κώδικα συμπεριφοράς που θα είναι πραγματικά άξιος να λέγεται κώδικας συμπεριφοράς και πρότεινε πέρα από τα άρθρα 14 και 15 και μια κοινή δήλωση μεταξύ Κοινοβουλίου και ε, Συμβουλίου το δεχτήκαμε αυτό, αλλά μόνο εάν μπει σε αυτή τη δήλωση πως τα κράτη-μέλη θα κινηθούν στο πνεύμα του κώδικα συμπεριφοράς όσον αφορά την σύνταξη των επιχειρησιακών προγραμμάτων και η Κομισιόν θα ε, υποβάλει το συντομότερο δυνατόν το τι θα περιέχει αυτός ο κώδικας. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Και το απόγευμα βέβαια θα ξανασυνεδριάσει η διαπραγματευτική ομάδα, αλλά αυτό το είχαμε ήδη συμφωνήσει και δεν δέχομαι συμφωνημένα κείμενα να αλλάζουν μόνο μονομερός. Δεν επιτρέπεται αυτό, το λέω ξεκάθαρα και ανοιχτά, γιατί ε, θα πρέπει να μας απασχολήσει ξανά το απόγευμα. Τώρα, Όσον αφορά το σπάσιμο σε δύο κομμάτια της ε, συμφωνίας ε, εταιρική ε, σχέσης που ανέφερε ο Λάμπερτ, εμείς είπαμε αρχικά πως φτάνει αρκεί να κάνουμε μια επαρκή συμφωνία. Γι' αυτό στο άρθρο 87 δεν είχαμε τόσο πολλές δυσκολίες για το σπάσιμο. Εντάξει, ήταν ζητήματα λεπτομεριών δύσκολα αλλά νομίζω πως ε, υπήρξε ένας αμοιβαίος συμβασμός που μας βοήθησε όλες τις πλευρές και βεβαίως ήταν δύσκολος αυτός ο διαχωρισμός όπως είπαμε. Εκεί πέρα είχαμε κάποια κομμάτια τα οποία το Συμβούλιο ήθελε να μπουν στο δεύτερο να μπουν από το δεύτερο κομμάτι στο πρώτο, γιατί ήταν, είχαν στρατηγική σημασία. Δηλαδή, ε, ρυθμίσεις για να υπάρξει συντονισμός μεταξύ κονδυλίων ε, του κοινωνικού ε, ταμείου και λοιπόν μείωση των διοικητικών δυσκολιών όλα αυτά ήθελα να μπουν στο πρώτο μέρος είναι ένας συμβιβασμός οπωσδήποτε, αλλά θεωρώ πως εμείς ως Κοινοβούλιο μπορούμε να το δεχτούμε και είχαμε πει στην Κομισιόν ε, πως ε, θα πρέπει να δει πως ε, θα μπορέσει να το ρυθμίσει για να είναι όντως ένας συμβασμός. Και έτσι τελικά συμφωνήσαμε στα άρθρα 14 και 15 όπως αυτά τροποποιήθηκαν. Στα υπόλοιπα άρθρα μπορεί να με συμπληρώσει ο Λάμπερτ, ε, υπήρχαν μικρές ε, αλλαγές. Κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι πως ε, είχαμε κοινή, κοινές διαπραγματεύσεις για το ότι χρειαζόμαστε πραγματικά ένα πλαίσιο διαφάνειας όσον αφορά την δημοσιότητα που ήταν δύσκολο για το Συμβούλιο αλλά σε διάφορα σημεία στο στρατηγικό προγραμματισμό ε, έγινε δεκτό και αυτό και αυτό είχε διαγραφεί πριν από τον, ε, μετά τον τελευταίο τριμερή διάλογο και αυτό πρέπει απόψε να δούμε ότι συμφωνεί με τα συμφωνημένα. Οπότε οι αλλαγέ οι οποίες έγιναν ε, πραγματικά ήταν θετικές, είναι κάποιες προσαρμογές και πρέπει να δούμε πώς ε, θα φροντίσουμε ως κοινοβούλιο το ότι ε, τα κράτη-μέλη διαφέρουν. Είναι άλλα με κεντρική διοίκηση, άλλα με ομοσπονδιακή δομή και πολλά με ενδιάμεση κατάσταση. Οπότε πρέπει να δούμε τις διαδικασίες που θα χρησιμοποιηθούν και έτσι τελικά νομίζω μπορούμε να πούμε πως εάν το εγκρίνουμε όπως το έχουμε συζητήσει, νομίζω πως έχουμε κάνει ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός και ε, πως θα έχουμε μια βάση και για τις ε, περιφέρειες μπορούν να ξεκινήσουν τον προγραμματισμό αλλά και για τον περαιτέρω τριμερή διάλογο. Μια παρατήρηση ακόμα. Το Συμβούλιο θα ήθελε να φύγουν αυτοί οι οριζόντιοι στόχοι. Εμείς ε, το υπερασπιστήκαμε και είπαμε πως ε, έχουμε και τη δημογραφική εξέλιξη, την ισότητα των ευκαιριών, ε, πρόσβαση για αναπήρους, ε, τις γυναίκες, αλλά και το, το θέμα των οικοσυστημάτων, της αηφόρου ανάπτυξης. Αυτά έμειναν μέσα, κάτι το οποίο επιθυμούσαμε ευθύς εξ αρχής και το Συμβούλιο δεν ήθελε καθόλου. Αλλά νομίζω πως ε, καταφέραμε να μείνει, να μείνει εντός και είναι αναγκαίο για τον προγραμματισμό. Ελπίζω να μην ξέχασα τίποτα. Λάμπερτ, θες εσύ? Όχι, όχι, δεν, δεν ξέχασες τίποτα, αλλά θέλω να πω το εξής. Ε, απόψε, θέλουμε αυτή τη μερική ε, συμφωνία και η πρότασή μου είναι η Κωνσταντσε να, να μιλήσει στη διαπραγμάτευση γιατί έχει έτσι τη σωστή, σωστή διάθεση να μην δεχτεί τίποτα προς λάθος ε, κατεύθυνση. Και είναι σημαντικό η εντολή ε, που μας δώσατε μας έδωσε τη δυνατότητα να πάμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και τώρα τα κονδύλια έχουν μια καλή ε, εξέλιξη και πρέπει βεβαίως να παραμείνει αυτή η επιτάχυνση και στο επόμενο κομμάτι της ε, θεματικής κέντρωσης του Κοινωνικού Ταμείου. Και να, να υπάρξει αυτή η πρόοδος. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε το, το καλύτερο αποτέλεσμα και τη σωστή, σωστή ταχύτητα. Και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που προσαρμόζονται όσον αφορά το πώς γίνονται οι αναθεωρήσεις, στο χρονοδιάγραμμα. Αλλά όταν το, το γράφουμε, ελπίζω να, τα καταφέρουμε, να, να δώσεις και εσύ τον αγώνα. Καλό είναι να, να δώσεις τον αγώνα απόψε για να στείλουμε τις πληροφορίες αμέσως στους συναδέλφους με όλα τα, τα άρθρα. Ναι, θα ήθελα τώρα να ρωτήσω τους κοιοδησηγητές. Ο Ήβαλς θέλει να πει κάτι. Ελίζ, Ελίζαμπεθ Σρέτερ. Ο Ήβαλς είναι ικανοποιημένος για την ώρα. Ναι, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα ως μια σιωπηλή παρατηρήτρια της διαπραγμάτευσης πρέπει να πω πως υπάρχει μια μέθοδος στην οποία καταλήξαμε τις τελευταίες 14 ε, ημέρες ε, η οποία για εμάς είναι απαράδεκτη. Το είπε η Κωνσταντς αλλά θεωρώ πως ε, είναι άδικο και απαράδεκτο μετά τις παραχωρήσεις που κάναμε στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο προσπαθεί, παρά το ότι κάποια πράγματα έχουν κλείσει, ε, να μας λέει πως λείπουν, παρά το ότι έχουν κλείσει. Δεν υπάρχει ακόμα το, το benchmark. Δεν ξέρω πόσες φορές το έχουμε πει. Μας υποβάλλει κείμενο το οποίο δεν συμφωνεί με αυτά που έχουμε αποφασίσει και συμφωνήσει. Συστηματικά δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ε, προσπαθεί να υπονομεύσει την θέση μας. Δεν γράφει αυτά τα οποία αποφασίσαμε. Έτσι λέει, ναι, μια διαφορετική διατύπωση, αλλά δεν είναι τεχνικό, είναι τελείως πολιτικό και αλλάζει το κείμενο. Και αυτό είναι ακριβώς στους τομείς που είναι για εμάς σημαντικοί και εμείς συμφωνήσαμε σε αυτό το διαχωρισμό για την συμφωνία εταιρική σχέση, το οποίο για μας δεν είναι καλή μέθοδος και εκεί πέρα όπου ακριβώς θεωρούμε πως πρέπει να επιτύχουμε κάποια πράγματα εκεί πέρα ακριβώς το υπονομεύουν τι να σου πω, από, από, από την Παρασκευή μέχρι σήμερα δηλαδή, τρει-τέσσερι φορέ, δεν μέτρησα πόσε φορέ το έκαναν, δεν είναι κατάσταση αυτή. 7 Δεκεμβρίου αποφασίσαμε τον κώδικα συμπεριφορά. Και το, το ξαναείδαμε. Μεταβλέπω το, το σημερινό κείμενο και δύο-τρία διαφορετικά κείμενα που προέκυψαν. Και εξακολουθεί να μην υπάρχει μέσα. και υποτίθεται πως ε, είχαμε μια κοινή δήλωση η οποία δεν, σημαίνει τίποτα τελικά. Εντάξει, καταλαβαίνω αυτό το οποίο φοβάται το Συμβούλιο. Φοβάται πως μετά η Κομισιόν θα μπει στα χωράφια της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης. Δεν ξέρω, ίσως μπορεί να μας εξηγήσει και η Κομισιόν. Δηλαδή, αν δεν πάει καλά η εταιρική σχέση... Ε, να φροντίσουν να το εξασφαλίσουν. Αλλά η μέθοδος την οποία ακολουθούν είναι πως ε, δεν θέλουμε οι εταίροι να συμμετέχουν στην προπαρασκευαστική φάση. Ε, μα δεν γίνεται αυτό. Γιατί όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται τώρα όσον αφορά τον προγραμματισμό μαζί με τους εταίρους. Και είναι σαφές πως σε όλες τις παραγράφους όπου μιλούσαμε για προγραμματισμό, όπου συζητήσαμε αυτά τα πράγματα, σε όλες ε, τις φάσεις, ε, λέγαμε εμείς, σε όλες τις φάσεις του ε, προγραμματισμού θα πρέπει να συμμετέχουν οι εταίροι. Και το σβήνανε συνέχεια. Και το λέγανε τεχνική διόρθωση ή νομική αναδιατύπωση, αλλά είναι ουσία. Έτσι αλλάζει ουσία. Δηλαδή ή, γράφουμε κάτι ή, ή γράφουμε ή δεν γράφουμε κάτι. Να αποφασίζουμε κάτι και μετά αλλάζουν το κείμενο. Ε, είναι απαράδεκτο. Και πρέπει να σας πω, ειλικρινά, εάν δεν ε, δω το αρχικό κείμενο, θα, θα έχω πρόβλημα. Να, να υποστηρίξω τον, ε, τον συμβασμό με το, με το Συμβούλιο. Το ανέφερε και η Κωνσταντσα. Πρέπει να έχουμε μια διάφανη διαδικασία για να γίνει μια δημόσια διαβούλευση. Απευθύναμε μια επιστολή λοιπόν, τα στοιχεία αυτά έχουν μπει μέσα στην εντολή μας και τα είχαμε διαπραγματευτεί και ξεκαθαρίσει. Και το Σαββατοκύριακο μας στέλνουν ένα κείμενο και τα έχουν σβήσει πάλι από μέσα. Δεν είναι, δεν είναι κατάσταση αυτή. Και πρέπει να σας πω, είναι σημαντικό ε, η Επιτροπή μας ε, να, να στηρίξει την εισηγήτρια και τη διαπραγματευτική ομάδα και πρέπει να τηρούνται οι συμφωνίες. Μπορεί έτσι να θέλει να κινείται το, το Συμβούλιο, αλλά δεν το δεχόμαστε, δεν είναι πράγματα αυτά. Βλάσεκ. Κύριε Βλάσεκ, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι από όλη αυτή την προσέγγιση αισθάνομαι ότι εμείς είμαστε ενωμένοι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και εκτιμώ βαθύτατα την εργασία της διαπραγματευτικής μας ομάδας. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει συμβιβασμός, δεν μπορούμε πάντα να βγαίνουμε κερδισμένοι. Έχω όμως εμπιστοσύνη και χαίρομαι που υπάρχει κυρίως εδώ ορισμός της αρχής που μας είναι τόσο προσφυλής, της εταιρικής σχέσης. Και αν συνεγγίσουμε την δική μας ε, προσέγγιση, ε, θα επιτύχουμε, δεν έχω να προσθέσω τίποτε. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Φτάνουμε σχεδόν στο τέλος του πρώτου μέρους των διαπραγματεύσεων και πιστεύω ότι μπορούμε ήδη να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Θα επιμείνω και συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη του συναδελφού Βλασάκ για την ε, ενότητα της ε, διαπραγματευτικής μας ομάδας. Προχωρούμε ενωμένοι, ενιαίοι και νομίζω ότι πρόκειται για σημαντικό στοιχείο. Κατορθώσαμε να ξεπεράσουμε τα πολιτικά συμφέροντα που πολλές φορές μας κάνουν να έχουμε αποκλίνουσες από στην Επιτροπή μας για να προχωρήσουμε ενωμένοι για να προσφέρουμε τα συμφέροντα των περιφερειών μας ε, μπροστά στους ε, άλλους εταίρους διαπραγμάτευσης. Πράγμα το οποίο προσδίδει ιδιαίτερη ισχύ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση. Παίρνουμε μένος σε αυτές τις διαπραγματεύσεις πεπισμένοι και αποφασισμένοι να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Δηλαδή, είμαστε πεπισμένοι ότι είμαστε σε διαπραγμάτευση. Δεν ισχύει βεβαίως το ίδιο, και αυτή ήταν και η αρχή θέση που εξέφρασε το Συμβούλιο, που είναι συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις και συνειδητοποιεί παρόλα αυτά σιγά σιγά ότι πρέπει πραγματικά να διαπραγματευτεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πράγμα το οποίο εξηγεί και την πρόοδο η οποία επιτεύχθηκε. Η αρχή της διαπραγμάτευσης είναι ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε τα πάντα και αμέσως. Υπάρχει όμως πρόεδρος όσον αφορά την σύμβαση εταιρική σχέσης, όσον αφορά το κώδικα συμπεριφοράς και ο απόψινός τριμερής διάλογος θα είναι σημαντικός. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι το 2013 θα πρέπει να ασχοληθούμε με πολύ σημαντικά θέματα για τα οποία έχει εκφράσει με απόλυτη σαφήνεια τη θέση η Επιτροπή μας. Το θέμα της ε, ε, μακροοικονομικού στόχου της οικονομικής και το θέμα των ε, θεματικών στόχων. Πιστεύω ότι στο πρώτο θέμα για το πρώτο θέμα θα πρέπει να λάβουμε εμείς θέση αποφασιστικής σημασίας σε σχέση με αυτά που λέει το Συμβούλιο, να εκφράσουμε ενωμένη την άποψή μας. Όσον αφορά τους θεματικούς στόχους, ελπίζω ότι θα κατορθώσουμε να ε, διατηρήσουμε τις ε, Αλλαγέ τι οποίε έχουμε επιφέρει στα έγγραφα τη Επιτροπή, όπω η προσία του περιβάλλοντο, η έννοια τη θέση ε, ε, απασχόληση ποιότητα, η ενίσχυση των ε, δυνατοτήτων που έχει κάθε εταίρος, πράγμα το οποίο πολλές φορές παραγνωρίζεται, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που θέλω να κάνω προς το παρόν. Σας ευχαριστώ. Ο Ιωαχήμ Τσέλερ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ακούω πως ε, βεβαίως επικρατεί δυσαρέσκεια για αυτά τα οποία ε, έχουν γίνει. Έχουν γίνει δέκα ε, διαπραγματεύσεις και αποτέλεσμα ελάχιστο. Μα άμα είμαστε τόσο εκνευρισμένοι, γιατί είμαστε τόσο ευγενικοί, ήμασταν τόσο ευγενικοί χτες. Χτες ε, ήταν εκεί πέρα το Συμβούλιο. Ήταν εδώ πέρα ο κύριος Μαυρογιάννης, ευγενέστατος, και έπρεπε να του τα πούμε αυτά τα πράγματα. Γιατί, έτσι όπως μου τα λέτε, η στρατηγική του Συμβουλίου είναι ξεκάθαρη χρονοτριβούν για να μην καταλήξουν πουθενά οι διαπραγματεύσεις. Και μετά να έρθουν και να μας πούνε «Α, φίλοι, τώρα πρέπει να αποφασίσουμε γρήγορα. Είτε συμφωνείτε, είτε φταίτε εσείς» για το ότι δεν θα εφαρμοστεί η πολιτική συνοχή. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει εμένα είναι τι ρόλο παίζει η Κομισιόν. Είναι τριμερής ο διάλογος. Η Κομισιόν είναι στο δικό μας το πλευρό, έκανε αυτό το οποίο έκανε πάντα. Δηλαδή τελικά πάει με τα κράτη-μέλη. Ήταν νομίζω οι εκπρόσωποι τη Κομισιόν στα κρατημέλη, στις περιφερειές και πρέπει να διορθώσω κάτι το οποίο είπα χτε. Γνωρίζω από κάποιους πως ε, σταμάτησε η επεξεργασία των επιχειρησιακών προγραμμάτων γιατί ελπίζουν πως θα ε, επέλθουν βελτιώσεις μέσω του Κοινοβουλίου. Αλλά Εν μεταξύ γνωρίζω από κάποια κράτη-μέλη και περιφέρειες πως έχουν δώσει εδώ και καιρό τα επιχειρησιακά τους ε, προγράμματα με βάση την πρόταση της Κομισιόν γιατί θεωρούν πως δεν θα αλλάξει και τίποτα σοβαρό και θα καταλήξουμε τελικά σε μια θέση η οποία δεν ε, θα αντικατοπτρίζει και τη συνθήκη της, ε, της Λισαβόνας. Δεν θα μπορεί δηλαδή να, να ακουστεί η φωνή μας στην διαμόρφωση των κανονισμών. Οπότε θα ήθελα να δώσω δύο λόγια για το τι έχει κάνει η Κομισιόν εδώ πέρα στην όλη αυτή διαπραγμάτευση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα σχόλια πριν δώσω ξανά τον λόγο στην Κωνσταντσε, Λαμπέρ και στην Κομισιόν. Για να Δεν συμπεριφερθήκαμε διαφορετικά χθε, Απλώ είμαστε πολύ πιο διπλωματικοί. Και είχαμε μια πολύ διπλωματική συζήτηση με την Προεδρία, αλλά νομίζω ότι μπόρεσαν να καταλάβουν τις επικρίσεις που κάναμε ή του Συμβουλίου. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο θέματα τα οποία πρέπει να ερωτηθούν. Ένα γενικό. Κάνω λάθος ή μας εξήγησε η νομική υπηρεσία της Επιτροπής και του Συμβουλίου ότι η συμβάσεις δεν μπορούν να γίνουν για θεσμικούς λόγους. Κάνω λάθος. Ο κύριος Βαν Ρομποϊ ετοιμάζει διαφορετικές συμβάσεις για τα διάφορα κρατημέλη ή... Τι αφορά αυτό το θέμα της συμβάσεις? Αυτή είναι η πρώτη γενική ερώτηση, αλλά δεν ξέρω σε ποιον την υποβάλλω. Ή είναι δυνατόν να γίνουν συμβάσει ή όχι. Συμβάσει συμβάσεις, όπω θέλετε. Δεύτερο θέμα, το περιεχόμενό τους. Την Άντια έχουμε κάτι διαφορετικό από τη συμβάση. Κατάλογος κριτηρίων, κατάλογος πόλεων και τώρα πρόταση του Συμβουλίου συμπεριλαμβάνει τις αρχές της προπαρασκευής. Δεν ξέρω αν υπήρχε το τελικό κείμενο για το θέμα το αστυνομικό. Υπάρχουν άλλα σχόλια από την Επιτροπή. Εάν όχι, ο κύριος Μπρόκερ, εκπρόσωπος της Επιτροπής. Thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποιες γενικές παρατηρήσεις να κάνω, εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάποιες παρατηρήσεις στη συνέχεια για πιο λεπτομερή ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν σήμερα. Ξεκινάοντας με την κατάσταση στα τέλη του 2012, βλέπουμε ότι υπήρχαν πάρα πολλές προκλήσεις στα πλαίσια της πρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τους έξι αυτούς κανονισμούς. Έχει σημειωθεί πολύ ικανοποιητική πρόοδος και βλέπουμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, δηλαδή τα τρία θεσμικά όργανα, συνειδητοποιούν ότι η κατάσταση πιέζει ιδιαίτερα, ότι είναι επίγουσα η κατάσταση. Και αυτό φάνηκε από την πολύ καλή πρόοδο που είχαμε και χθε, αλλά και στου υπόλοιπου τομεί. Είδαμε ότι για τους περισσότερους τομείς είχαμε τριμερείς διαλόγους οι οποίοι σημείωσαν σημαντική πρόοδο. Και βέβαια έχουμε και συγκεκριμένε διατάξεις όσον αφορά τα στρατηγικά προγράμματα και το CPR. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει σιγά σιγά μια πρόοδος που θα μας οδηγήσει σε συμφωνία στο τέλος. Καταδεικνύουν όλα αυτά την δέσμευση και τις προσπάθειες τόσο του εισηγητή όσο και των σκιωδών εισηγητών και χάρη στη δική του συμβολή καταφέραμε να έχουμε αυτή τη σημαντική πρόοδο. Τώρα, όσον αφορά το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελπίζω να θεωρείτε κι εσεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατήρησε επικοδομητικό ρόλο. Αυτή ήταν η αρχική μα πρόθεση. Προφανώ, εμεί υπερασπιστήκαμε την πρότασή μα στα σημεία αυτά που θεωρούσαμε ότι έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο και κάθε φορά αιτιολογούσαμε τη στάση μα. Βέβαια, σεβαστήκαμε απολύτω και τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ω συνομοθέτη που συμμετέχει αυτή τη στιγμή με μια διαφορετική νομοθετική διαδικασία από ό,τι στο παρελθόν. Δεν μπορούμε εμεί να μένουμε στη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν βλέπουμε ότι δεν υποστηρίζεται από του νομοθέτε. Επίση, προσπαθήσαμε να είμαστε επικοδομητικοί, ψάχνοντα συμβιβασμού μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και πολλές φορές κάναμε κάποιες ε, ουσιαστικές προτάσεις στη δικασία της σύνταξης των εγγράφων για να καταλήξουμε τελικά σε ένα συμβιβασμό. Επίσης, ε, επικεντρωθήκαμε στην νομοθεσία καλής ποιότητος. Είπαμε ότι θέλουμε να καταλήξουμε σε κανονισμούς οι οποίοι να λειτουργούν στην πράξη, πραγματικά να δημιουργούν ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να μην είναι θεωρητικό, αλλά να μπορεί να αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για τα κράτη-μέλη, τις περιφέρειες, τις τοπικές αρχές, προκειμένου να καταφέρουν να εφαρμόσουν επιτόπου προγράμματα και να μπορούν οι δικαιώχοι να αποφεληθούν από τα προγράμματα αυτά. Αυτό είναι από τους σημαντικούς ρόλους που διδραματίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να έχουμε δηλαδή ένα, μια πολύ καλή ποιότητα στο τελικό αποτέλεσμα. Τι σημαίνει όμως τώρα αυτό για τα ιδιαίτερα σημεία του στρατηγικού προγραμματισμού. τα οποία αποτελούν τμήμα της πολύ μεγάλης προσπάθειας που έγινε τις τελευταίες εβδομάδες ανάμεσα στα θεσμικά όργανα. Προφανώς θέλουμε να πετύχουμε μια συμφωνία για τα σημαντικά αυτά νομοθετήματα. Για τη συμφωνία αυτή πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσει την απαραίτητη βάση, ένα νομικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να αρχίσουν να προετοιμάζουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα. Αυτό είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύουμε ότι θα κινητοποιήσει θετικά και τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις που θέλουμε να γίνουν προκειμένου να τηρήσουμε το αρχικό μας χρονοδιάγραμμα. Τι προτάθηκε τώρα για τη συμφωνία εταιρική σχέση. Δεν ήμασταν υπέρ του διαχωρισμού, αλλά θεωρούμε ότι ο συμβασμό στον οποίο καταλήξαμε είναι τελικά καλό και εν γέννη πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει ο συμβασμός αυτός να πετύχουμε ένα συμβασμό και για τον κώδικα συμπεριφοράς. Η συμφωνία λοιπόν που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας θεωρούμε ότι είναι θετική, αλλά όπως υπόθηκε πολλές φορές, ο διάλογος κρύβεται πάρα πολλές φορές στις λεπτομέρειες. Τις τελευταίες ημέρες αναφερθήκαμε σε επιμέρους σημεία των κανονισμών είπαμε ότι δεν θα πρέπει να επέλθουν αλλαγέ σε κάποιες λεπτομέρειες του κανονισμού που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα. Είτε για τη διατήρηση των βασικών ενιών του κώδικα συμπεριφοράς, είτε προβλήματα τα οποία θα δημιουργούσαν κάποια βεβαιότητα ή για κάποιες μελλοντικές διεργασίες, για την μελλοντική εφαρμογή αυτών των κανονισμών. Όσον αφορά την ε, αναδρομική εφαρμογή του κώδικα συμπεριφοράς, αναφέρθηκε και αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ο κώδικας συμπεριφοράς που θα αρχίσει να ισχύει μετά την έγκριση της βασικής πράξης δεν μπορεί να έχει αναδρομική φύση. Λέμε λοιπόν ότι τα όσα λέγονται στον κώδικα συμπεριφοράς δεν μπορούν να ισχύσουν αναδρομικά έτσι ώστε να μπλοκαριστεί η έγκριση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης. Αυτό λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε και μία δήλωση η οποία θα πηγαίνει σε αυτή την κατεύθυνση. Πέρα όμω τώρα από τον κώδικα συμπεριφορά υπάρχουν και άλλα σημαντικά σημεία στο ίδιο το άρθρο 5, στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο. στοιχεία τα οποία θα πρέπει να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη και τα οποία θα πρέπει να, στα οποία θα πρέπει να δώσουμε τη δέουσα σημασία. Μία τελευταία παρατήρηση όσον αφορά την ονομασία που θα δοθεί σε αυτές τις συμφωνίες εταιρική σχέση. Εμείς δεν είχαμε τοποθετηθεί πάρα πολύ ισχυρά ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είχαμε καταλήξει σε κάποια τοποθέτηση. Είχαμε απλώς πει ότι η εταιρική αυτή σχέση, η συμφωνία εταιρική σχέσης θα πρέπει να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι λοιπόν ένα έγγραφο το οποίο υπογράφουν τα δύο συμβαλόμενα μέρη όπως γίνεται συνήθως. Αυτή τη διαφοροποίηση θα ήθελα να κάνω σε σχέση με τις συμβάσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Όλμπρεχτ. Οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται σε διαφορετικό πλαίσιο και με διαφορετικό τρόπο. Έχουμε βέβαια κάποιες ανησυχίες ότι προσπαθώντας να καταλήξουμε σε μια γενική συμφωνία, εκκρεμούν ακόμα κάποια ζητήματα, ζητήματα επί των οποίων πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις και διορθώσεις. Πιστεύω όμως ότι θα γίνει και αυτό και στηρίζομαι και στην δική σας υποστήριξη προκειμένου να καταφέρουμε να κάνουμε αυτές τις βελτιώσεις. Σας υπενθυμίζω τα κράτη-μέλη χρειάζονται αυτή την νομοθετική βάση για να λειτουργήσουν. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Κωνσταντσε. Ναι, για να κλείσω κάποιες παρατηρήσεις ε, το θέμα της σύμβασης, η συμφωνίας, ε, ρωτήσαμε και την νομική μας υπηρεσία η οποία λέει και τα δύο είναι νομικά δεσμευτικά και σημασία έχει το περιεχόμενο της ε, συμφωνίας και όχι το όνομα. Γιατί δεν ήθελε να αποκλίνει η Πρόεδρια και ήθελε να μείνουμε στη συμφωνία. Βεβαίω αυτό κοστίζει και στο Συμβούλιο, γιατί είπαμε πως ε, εντάξει θα το δεχτούμε, αν δεχτεί το, το Συμβούλιο τη Σύμβαση. Τώρα απόψε θα ξεκαθαρίσουμε τι θα γίνει. Το ερώτημα γιατί χτες ε, ήμασταν τόσο ευγενικοί. Μα με ξέρετε όλοι, μπορώ να είμαι ε, πάρα πολύ έντονα. Χτες προσπάθησα να είμαι φιλική, γιατί δεν διαπραγματευτήκαμε με τον Υπουργό ε, με τον συναδελφό του, τον, ε, τον Αντώνη. Και χτες ε, ήρθε εδώ πέρα για να κλείσει την Προεδρία και επιτύχαμε αρκετά. Δεν θέλω να το υποβιβάσω. Είναι ένα στρατηγικό κομμάτι του γενικού κανονισμού, στο οποίο επιτύχαμε συμβιβασμούς και στην αρχή των διαπραγματεύσεων δεν πίστευα ποτέ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, ότι θα έρθει τόσο πολύ με το, μέρο μας, με το μέρος μας στο Συμβούλιο, ούτε ότι θα δεχτεί τον κώδικα συμπεριφοράς, ε, την ε, προσέγγιση των πολλών ταμείων, την οριζόντια πτυχή. Πάρα πολλά στοιχεία τα οποία περάσαμε. Και άρα μπορούσαμε χτες να πούμε ε, ικανοποιημένοι πως είναι εντάξει κάποια στοιχεία, ε, χρειαζόμαστε και την κάλυψη της Επιτροπής γιατί συνεχίζεται ακόμα ο τριμερής ε, διάλογος ε, και πρέπει να μας στηρίξετε στην εντολή μας και να πούμε πως ε, πρέπει απόψε να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά στην διαπραγμάτευση για να προχωρήσουμε λίγο ακόμα προς σωστή κατεύθυνση. Ε, οπωσδήποτε υποθέτω πως απόψε θα έχουμε μια συμφωνία, αλλά πρέπει και επιτέλους το Συμβούλιο να γράψει αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει στη συμφωνία. Γι' αυτό χτες ήμουν έτσι κάπως διπλωματική, ε, αλλά πρέπει να μιλάμε καθαρά, γιατί αλλιώς θα χάσουμε τη διαφάνεια που ε, είχαμε επιτύχει. Και ε, εάν το χάσουμε αυτό θα είναι δύσκολες οι διαπραγματεύσεις στο μέλλον γιατί πρέπει και οι συνάδελφοι να μπορούν να βασιστούν πως ε, είμαστε εντός της εντολής που μας έχουν δώσει. Ευχαριστώ. Jan, you are biting into your time for your report, so, but you are allowed. Αν τρως χρόνο από τη δική σου έκθεση, αλλά έχεις το λόγο. Yes, Chair, exactly. You have, ναι, ναι, ναι. Σωστά τα λες, Πρόεδρε. Θα ήθελα να προτείνω κάτι ο συναδέλφους στην διαπραγματευτική ομάδα. Είναι κάπως ασαφή τα πράγματα. Το ερώτημά μου είναι, υπάρχει συμφωνία της συμβάσης. Η νομική υπηρεσία είπε ότι δεν μπορούμε να έχουμε σύμβαση μεταξύ κομισιών και κρατών μελών. Αλλά δεν υπάρχει και τίποτα μεταξύ κρατών μελών και επιτροπής. Το ερώτημα λοιπόν είναι, ή σε εθνικό επίπεδο έχουμε συμφωνία μεταξύ των εταίρων ή σύμβαση μεταξύ των εταίρων. Μετά τα πράγματα πάνε στην Επιτροπή, η οποία πρέπει να επαληθεύσει αν όλα αυτά έχουν γίνει σύμφωνα με τα νομι... τις νομικές πράξεις. Παρακαλώ, νομοθετικές πράξεις. Παρακαλώ λοιπόν, διευκρινίστε το αυτό. Υπάρχει συμφωνία μεταξύ Κομισιόν και κράτου μέλους ή συμφωνία μεταξύ εταίρων σε μία χώρα και μετά εγκρίνει αυτή τη συμφωνία η Κομισιόν. Εάν ο κώδικας συμπεριφοράς ε, συμφωνηθεί μεταξύ εταίρων της ιδίας χώρας ή μεταξύ χώρας εταίρων δηλαδή και κομισιόν είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Διευκρινίστε το αυτό. Το ρώτησα εγώ πριν από ένα χρόνο. Στην... Ποιοι είναι οι εταίροι. Οι εταίροι για μένα είναι στο εθνικό επίπεδο και υπάρχει συμφωνία σε εθνικό επίπεδο. Κάνω λάθος. Ίσως κάνω λάθος. Η Κωνσταντζα. Η σύμβαση εταιρική σχέσης που λέμε τώρα αν είναι σύμβαση ή συμφωνία είναι μεταξύ κράτους μέλους και κομισιών. Και εκεί πέρα προφανώς αγγλικά είναι αδιάφορο το εάν πούμε agreement είναι η contract είναι εξίσου νομικά δεσμευτικά. Το συζητήσαμε αυτό επί μακρόν. Στα γερμανικά δεν είναι το ίδιο. Γι' αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το θέμα αυτό. Το... Ε, έχουν συνεννοηθεί και οι νομικές υπηρεσίες των ε, θεσμικών οργάνων, αλλά είναι συμφωνία μεταξύ Κομισιών και κράτους μέλους. Στο εθνικό επίπεδο, αρχικά, στο άρθρο 5, είχαμε την προσέγγιση να γίνει μια συμφωνία μεταξύ εταίρων και κράτους μέλους. Αυτό δεν το περάσαμε στις διαπραγματεύσεις, αλλά συμφωνήθηκε να υπάρξει μια εταιρική σχέση, διόρθωσε με Λάμπερτ, όσον αφορά την κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, ε, την ε, εκτέλεσή τους, ε, τη διαχείριση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο. Όλα τα επίπεδα της δουλειάς δηλαδή όπου συμμετέχουν εταίροι. Αυτό είναι στο εθνικό επίπεδο και αυτό το καταφέραμε, αλλά η αρχή αυτή της εταιρική σχέσης στο εθνικό επίπεδο δεν είναι θέμα που πρέπει να αξιολογήσει πάλι η Κομισιόν, εκτός εάν είναι πράγματα τα οποία έχουν συμφωνηθεί στη Συμφωνία εταιρική Σχέσης. Οπότε έχουμε αφενός τη συμφωνία αυτή και λέμε πως είναι στρατηγικά σημαντικό το τι πρέπει να, να μπει εκεί πέρα μεταξύ κράτους μέλους και Κομισιόν και βεβαίως χρειάζεται άλλη ευελιξία για τις περιφέρειες. Ε, έχουμε την ευελιξία σε επιχειρησιακά προγράμματα, ε, συμφωνήσαμε γιατί είναι λογικό πάντα βεβαίως υπό πως θα τηρηθεί αυτή η αρχή της εταιρικής σχέσης στα κράτη-μέλη. Ε, μα δεν με ακούς άμα μιλάς. Στα κράτη-μέλη, στα κράτη-μέλη, φαίνεται. Το διαβάζετε αυτό στο άρθρο 5. Οι εταίροι είναι τοπικοί και περιφερειακοί. Ε, οι δημόσιοι φορείς, οι κοινωνικοί και οικονομικοί, μεγάλοι οργανισμοί. Στο άρθρο 5 υπάρχει ένας κατάλογος του τι, ποιος είναι εταίρος και σε ολόκληρο τον ε, συμβιβασμό παραπέμπουμε στα άρθρα 5, 7 και 8 όπου ε, υπάρχει η αρχή της εταιρική σχέσης και περιγράφεται και η διαδικασία. Ναι, στην κυβέρνηση. Και μετά η κυβέρνηση είναι ο εταίρος της Κομισιόν. Να ρωτήσουμε το, το, τον Διευθυντή της Κομισιόν να μας εξηγήσει. Ο Γιώχιμ Τσέλερ θέλει να μιλήσει. There is cost also to of this discussion. Ε, συνάδελφοι, όμως η συζήτηση τραβάει πολύ. Ναι, ναι, μα συνάδελφοι, αυτό ήταν ξεκάθαρο από πριν πως ε, η Κομισιόν θα συνάψει μία σύμβαση με τα κράτη-μέλη για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται εκεί. Το ένα ήταν αυτό. Και το άλλο, είχαμε τους εκπροσώπους, ακούσαμε τους εκπροσώπους των ΜΚΟ ότι εμείς θα έπρεπε να επιμείνουμε όταν κλείνουν αυτές οι συμφωνίες με δεσμευτικούς στόχους μεταξύ Κομισιών και κρατών μελών, να έχουμε φροντίσει το κράτος μέλος να ονομάσει τους εταίρους του και να δεσμευτεί νομικά και να έχουν το δικαίωμα ε, να επηρεάζουν τις αποφάσεις. Ε, αυτό δεν το ακούσαμε. Ακούσαμε από κάποιες περιφέρειες πώς τα συμβαλώμενα μέρη από πλευράς του Συμβουλίου δεν το σκέφτονται καν να συμπεριλάβουν με χαρακτήρα νομικό δεσμευτικό στις συμβάσεις τους εταίρους. Ναι, εντάξει, θα παρακολουθούν στις επιτροπές όσον αφορά την κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, αλλά όχι να συναποφασίζουν ε, για την επίτευξη των στόχων. Αυτό απορρίφθηκε. Εμάς στη Γερμανία. Τα κρατήδια είναι οι εταίροι και καταρτίζουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα. Έχουν επίσης δική τους καθορισμένη θέση συνταγματική, ε, αλλά αυτό δεν ισχύει για τις περισσότερες περιφέρειες ε, της Ευρώπης που έχουν σαφώς ε, υποδέστερη θέση έναντι του κράτους μέλους. Και ξέρω ήδη κάποια κράτη-μέλη τα οποία έχουν φτιάξει τα επιχειρησιακά τους προγράμματα και δεν σκέφτονται να εμπλέξουν ε, περιφέρειες λοιπά. Παρά το ότι μιλάμε για αστική διάσταση, ε, πέρα πρέπει να, να μπούμε στη συζήτηση και να ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν θέλει να, να μπει στη συζήτηση αυτή. Κύριε Πρόεδρε, ε, Πρόεδρος Διακόπτη, να ολοκληρώσουμε και γρήγορα όμως. Ναι, θα είμαι σύντομος. Η Συμφωνία Εταιρική σχέση είναι συμφωνία ανάμεσα στο κράτο μέλο και την Επιτροπή. Συμφωνία που θέτει τι προτεραιότητε χρηματοδότηση για το σύνολο του κράτου μέλου, του αναφέρει του θεματικούς στόχους που θα επικεντρωθεί, στου οποίου θα επικεντρωθεί το κράτο μέλο και αναφέρεται επίση και στον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν οι οριζόντιε αρχέ, ο τρόπο με τον οποίο θα γίνει ο συντονισμό με άλλου μηχανισμού χρηματοδότηση και άλλα ταμεία. Πρόκειται δηλαδή για μια συμφωνία ανάμεσα στο κράτο μέλο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στι αρχέ τώρα αυτέ τη εταιρική σχέση προβλέπεται ο τρόπο με τον οποίο το κράτο μέλο θα εφαρμόσει το πρόγραμμα το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Και εδώ πέρα έχουμε τη συμμετοχή των τοπικών αρχών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, θα πρέπει να συμμετέχουν και αυτοί στη διαδικασία στο πλαίσιο του κράτους μέλους για την προετοιμασία και την εφαρμογή της εταιρικής σχέσης και για την εφαρμογή κάθε επιμέρους προγράμματος και όλες τις λεπτομέρειες για το πώς θα πρέπει να οργανωθεί αυτή η εφαρμογή, αυτό, σε αυτό ουσιαστικά επικεντρώνεται ο κώδικας συμπεριφοράς. Πώς θα ισχύσει επιτόπου η εταιρική σχέση. Λαμπέρτ, πάλι σας να μιλήσει με σχέση που πριν από λίγο ότι κουράστηκε. Ναι, ναι, αλλά πρέπει να διευκρινίσω κάποια πράγματα πρώτα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι ε, στέλνουμε εδώ πέρα διαφορετικά μηνύματα και αναφερόμαστε στις διαφορετικές έννοιες όσον αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αρχικά εγώ είχα την εντύπωση ότι το Συμβούλιο ήθελε ό,τι είχαν διαπραγματευτεί να συμπεριληφθεί 100% στο τελικό κείμενο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πάρα πολύ διστακτική τους τελευταίους μήνες και είδαμε βέβαια ότι όταν δυσκόλευαν τα πράγματα έκανε κάποιες συμβαστικές προτάσεις, το οποίο ήταν ιδιαίτερα θετικό. Οι διευκρινήσεις πάντως αυτές που μας δόθηκαν τώρα είναι θετικές. Εμείς στο δικό μας κείμενο είχαμε προτείνει συγκεκριμένα στο άρθρο 5 να έχουμε μία συμφωνία εταιρική σχέση, έτσι το ονομάζαμε, όπου θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους αυτούς τους αποκεντρωμένους φορείς να συμμετέχουν. Τώρα όμως από ό,τι φαίνεται δεν δίνεται τόσο πολύ αυτή η δυνατότητα. Δεν υπάρχουν τα κείμενα αυτά τα οποία θέλαμε εμείς, τα οποία προστάτευαν περισσότερο ή προωθούσαν τη συμμετοχή των περιφερειακών φορέων. Τώρα στο άρθρο 5 έχουμε θέσει πολύ συγκεκριμένε διατάξεις. Πρέπει να δούμε όμως πώς θα λειτουργήσουν στην πράξη τα πράγματα, τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Και θέλουμε τελικά να προωθήσουμε ένα θετικό κείμενο. Αυτό ελπίζουμε ότι θα είναι και έκβαση της ε, βραδινής συζήτησης που θα έχουμε σήμερα. Ο Γιάννο Ολμπρίχτ έθεσε ένα ερώτημα όσον αφορά τις αστικές περιοχές. Υπάρχει πλέον μια συγκεκριμένη εντολή που περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Εταιρική Σχέση και λέμε ότι η βασική αρχή για να εντοπίσουμε τι αστικέ περιοχέ όπου θα προβλέπεται δράση υποστήριξή του θα εντοπίσετε μέσα σε αυτή τη συμφωνία. Δεν δημιουργήσαμε ξεχωριστούς καταλόγους δηλαδή. Έχουμε εντάξει και την αστική διάσταση, τι αστικέ περιοχέ στην ενιαία αυτή συμφωνία εταιρική σχέσης. Και πραγματικά αισιοδοξώ ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα σήμερα το βράδυ. Θα είναι δύσκολο βέβαια, αλλά θα δούμε. Προεδρο, ευχαριστούμε λοιπόν. Ολοκληρώνουμε το σημείο αυτό. Σας ευχαριστώ όλου. Έχουμε ακόμα δύο σημεία στην ημερήσια διάταξη. Πρωτού τα καλύψουμε, να σας ενημερώσω για τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τους πολιτικούς συντονιστές χθε το βράδυ όσον αφορά τις ε, γνωμοδοτήσεις και μη νομοθετικές γνωμοδοτήσεις. Cultural Creative Sectors, ECR, θαλάσσιες μεταφορές και σχετικές πολιτικές, ΕΛΚΑ, επαναβιομηχανοποίηση της Ευρώπης, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Επίσης, συζητήσαμε εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας. Δύο αποφάσεις ελήφθησαν, μία για πρόταση του ΕΛΚΑ να συνταχθεί έκθεση ιδίες πρωτοβουλίας όσον αφορά τις επιπτώσεις των ε, δημοσιονομικών περικοπών για τις περιφέρειες και οι σοσιαλιστές πρότειναν έκθεση ιδίες πρωτοβουλίας όσον αφορά την ε, ενεργειακή αποδοτικότητα με έμφαση στην στέγαση. Επίσης, οι πράσινοι και οι γκούε θα υποβάλουν με γραπτή μορφή προτάσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν προφορικά μόνο χθε. Όσον αφορά τις εξωτερικές μελέτες, αποφασίστηκε να ζητήσουμε μία μελέτη από εξωτερικούς φορείς όσον αφορά την αξιολόγηση και την εφαρμογή των αρχών της εταιρική ε, σχέσης στα πλαίσια του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου. Θα πρέπει ενδεχομένως να αναδιατυπώσουμε λίγο το όνομα αυτής της μελέτης, την ομασία αυτής της μελέτης. Επίσης, οι συντονιστές θα πρέπει να αποφασίσουν για τις συγκεκριμένε ημερομηνίες των αντιπροσωπιών μας για το 2013, γιατί είχαμε αποφασίσει στο παρελθόν πού θα πάμε και ποιες εβδομάδες, αλλά τώρα πρέπει να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για ημέρες. Και έχουμε και δύο ακόμα εκθέσεις θα μας ενημερώσει καταρχάς ο Γιάνν Όλμπριχτ για τις ειδικέ διατάξεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και συνέχεια ο Βίκτορ Μποστινάρου θα μας ενημερώσει για το Ταμείο Συνοχής και για το πώς εξελίσσονται οι σχετικές διαπραγματεύσεις. Πρέπει μέσα στα επόμενα 20 λεπτά να καλύψετε και τα δύο αυτά σημεία. Δίνω καταρχάς το λόγο στον Γιάννα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάξτε, οτιδήποτε αποφασίσουμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ουσιαστικά εξαρτάται από το CPR. Είναι πάρα πολύ σημαντικός λοιπόν ο σημερινός τριμερής διάλογος και θα πειράσει βέβαια και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα είμαι σύντομος. Στον πρώτο τριμερή διάλογο συμφωνήσαμε για το πεδίο εφαρμογής των δράσεων, καθώς επίσης και για την αστική και δαφική διάσταση. Αυτά σα τα εξήγησα όμως ήδη. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή την τέταρτη στήλη από το Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίμασε τη δική της την εκδοχή. Περιμένουμε την τελική εκδοχή, την τελική στήλη από το Συμβούλιο. Στην δεύτερη συνάντηση που έγινε για τη θεματική συγκέντρωση, το Συμβούλιο δεν ήθελε να κλείσει κανένα κεφάλαιο προτού ληφθεί πρώτη τελική απόφαση για το CPR, και προτού ληφθεί και μία απόφαση ενδεχομένω για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί στα πλαίσια της θεματικής συγκέντρωσης έχουμε το πρόβλημα της ε, κατηγοριοποίησης των περιφερειών, ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα και για μας. Αναφέρομαι στις μεταβατικές αυτές περιφέρειες, γιατί από τη μια έχουμε τις πιο ανεπτυγμένες, τις λιγότερο ανεπτυγμένες, και υπάρχει έπειτα και στη συνέχεια η κατηγορία των περιφερειών αυτών που βρίσκονται ανάμεσα στις δύο αυτές κατηγορίες. Στην τελευταία πρόταση που έγινε στα πλαίσια του, δι... του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου περιλαμβάνονται και αυτές οι μεταβατικές περιφέρειες. Φαντάζομαι λοιπόν ότι στην τελευταία πρόταση που θα γίνει θα εγκριθούν από τα κράτη-μέλη και αυτές οι περιφέρειες. Αλλά το θέμα είναι πόσες περιφέρειες τελικά θα έχουμε σε αυτή την κατηγορία και τι αντιμετώπιση θα έχουν οι περιφέρειες αυτές όσον αφορά το ζήτημα της επιλεξιμότητας. Αυτό το οποίο εμείς προτείναμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να έχουμε τριών νηδών περιφέρειες, λιγότερο αναπτυγμένες, μεταβατικές και αναπτυγμένες. Δεν συζητήσαμε για χρήματα, δεν ήταν αυτό το δικό μας πρόβλημα, απλώς είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποιημένη θεματική συγκέντρωση και προτείναμε και τρεις κατηγορίες θεματικής συγκέντρωσης και όχι δύο όπως είχε πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν οι αναπτυγμένες και μεταβατικές περιφέρειες να μπουν στην ίδια κατηγορία, να έχουν την ίδια αντιμετώπιση, ενώ εμείς λέμε ότι πρέπει να έχουν διαφοροποιημένη αντιμετώπιση. Θεματική συγκέντρωση 50% για παράδειγμα στις λιγότερο αναπτυγμένες, 80% στις πιο αναπτυγμένες, ενώ εμείς προτείναμε 60% συγκέντρωση για τις μεταβατικές περιφέρειες. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν 80% οι αναπτυγμένες και οι μεταβατικές μαζί. και πιστεύουμε ότι τρεις, ότι τρεις θεματικοί στόχοι θα πρέπει να γίνουν τέσσερις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις τελευταίες διαπραγματεύσεις είπε ενδεχομένω ότι θα μπορούσε ο τέταρτος θεματικός τομέας να είναι το ICT, Information Communication Technology. Εμείς ε, είπαμε να μείνει ανοιχτός ο τέταρτος θεματικός τομέας και ακούσαμε σήμερα κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις μας είπαν ότι ενδεχομένω αν ο τέταρτος αυτός τομέας είναι οι μεταφορές, τότε δεχομένως να απορροφήσει πάρα πολλούς σπόρους από τους άλλους θεματικούς τομείς. Η συζήτηση λοιπόν που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι να μείνει ανοιχτό ο τέταρτος θεματικός τομέας ή να εγκρίνουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο τέταρτος θεματικός τομέας να είναι το ICT. Έχουμε επίσης και το ζήτημα του phasing out, της ε, βαθμιαίας μείωσης αν δεν υπάρχουν οι μεταβατικές περιφέρειες, τότε εμφανίζεται και αυτή η αρχή του phasing out. Αν υπάρχουν όμως οι μεταβατικές περιφέρειες, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Είπαμε ότι δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε επιπλέον κατηγορίες. Οι περιφέρειες που βρίσκονται στη φάση του phasing out να μπορούν να μπουν στην κατηγορία των μεταβατικών περιφερειών. Άλλες προτάσεις που γίνουν από τα κράτη-μέλη ήταν οι περιφέρειες της κατηγορίας phasing out να εξομοιωθούν ουσιαστικά με τις αναπτυγμένες περιφέρειες. Έχουμε επίσης πρόβλημα και με το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας, μάλλον όχι πρόβλημα γιατί οι περισσότεροι μάλλον θέλουν να αυξηθούν τα ποσοστά τα οποία έχουμε Επομένω, δεν υπάρχουν εδώ πέρα σημαντικά προβλήματα. Να αυξηθεί δηλαδή η χρηματοδότηση και για τι πιο αναπτυγμένε περιφέρειε όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα. Το πρόβλημα επίση έγκυται και στο τι θα κάνουμε με τι ε, άκρω αποκεντρωμένε περιφέρειε. Εδώ πέρα ακόμα δεν έχουν καταλήξει τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο. Εμεί δεν έχουμε μπλακεί πάρα πολύ στη συζήτηση αυτή. Πάντω αυτή είναι η συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη τουλάχιστον στο Συμβούλιο όσον αφορά τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι εμείς περιμένουμε την τέταρτη στήλη από το Συμβούλιο για το πεδίο εφαρμογής και δράσης και για τις αστικές περιοχές και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη θεματική συγκέντρωση όσον αφορά το CPR και όσο δεν ολοκληρώνται οι σχετικές συζητήσεις, δεν νομίζω το Συμβούλιο θα θελήσει να ανοίξει τη συζήτηση γι' αυτό. και θα συμφωνήσω και με την Κωνσταντς ολοκληρώνοντας, λέγοντας ότι ελπίζω και εγώ ότι οι Ιρλανδοί θα είναι όσο ικανοί είναι και ο Αντώνης. Όχι για τη μέθοδο εργασίας αναγκαστικά που δεν μπορεί να είναι η ίδια, αλλά πρέπει να πούμε ότι διατήρησε μια πάρα πολύ επαγγελματική στάση, είχε πολύ καλές γνώσεις, αλλά πολλές φορές ο τρόπος εργασίας ήταν λίγο προβληματικός. Πάντως πρέπει να αναγνωρίσουμε πραγματικά τα υψηλά επαγγελματικά πρότυπα τα οποία είχε η Κυπριακή Προεδρία. Πρόεδρος. Υπάρχει ένα λεπτό για σχόλια στην έκθεση αν θέλει κανείς να πει κάτι, αλλά κανείς δεν θέλει. Η Κομισιόν δεν έχει να προσθέσει τίποτα. Περνάμε λοιπόν στον Βίκτορα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Due to the fact that the council. Είχαμε μόνο μία συνάντηση, δεδομένου ότι έφτασε πολύ αργά με πρόταση το Συμβούλιο. Αλλά για τις εξελίξεις θα πω το εξής. Θα ευχαριστήσω την Κομισιόν για τη διαθεσιμότητά της. Είχαμε μια πολύ καλή προπαρασκευαστική συνεδρίαση πριν αρχίσει ο τριμερής διάλογος, πράγμα που οποίο βοήθησε πάρα πολύ τις προσπάθειες που είχαμε καταβάλει και εμείς για να καταλήξουμε σε αποτελέσματα. Τώρα όσον αφορά το ίδιο το περιεχόμενο του τριμερούς διαλόγου. Πρέπει να πω ότι γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένο με το αποτέλεσμα, διότι με τις διαπραγματεύσεις που δεν ήταν πολύ δύσκολες, Επιτύχαμε καλά αποτελέσματα. Τα πιο σημαντικά στοιχεία θα ήθελα να σας τα φέρω συνοπτικά. Τα κύρια σημεία στη συζήτηση ήταν επενδύσεις το περιβάλλον. Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για να συμπεριληφθεί το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ενεργειακή αποδοτικότητα και η μείωση των εκπομπών. Στο άρθρο 2 θέλουμε να γίνει αναφορά και στην ε, ε για κονδύλια που θα πίνουν από το Ταμείο Συνοχή. Η συμβουλή ήταν αντίθετο, μας είπε ότι η δεν έχει τέτοιου εντολή, αλλά εμείς επιμείναμε εκ μέρους της Επιτροπής με την εντολή που έχουμε από τον προηγούμενο Ιούλιο και είπαμε ότι στον κανονισμό του Ταμείου Συνοχής θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα θέματα εφόσον επηρεάζονται από τον κανονισμό. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία γιατί αυτό είναι σημαντικό, με την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποκλείσαμε όχι μόνο τον decommissioning, αλλά και την ε, δημιουργία νέων ε, πυρηνικών εργοστασίων. Και είχαμε την ίδια τροπολογία με το Συμβούλιο. Τι σημαίνει αυτό. ότι για τα θέματα τα ενεργειακά έχουν την ίδια θέση με ε, προηγουμένως για κάποια εργοστάσια ισχύως 20 ΜΒ. Επίσης, τα πλαίσια των προτεραιοτήτων επενδύσεων, φερθήκαμε στο άρθρο 3. Τελικά, χρησιμοποίηση ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, στέγαση και ανεργειακή απόδοση είχαμε την ίδια θέση ε, σχεδόν με το Συμβούλιο. Άρθρο 3. Προτεραιότητε επενδύσεων. Το Συμβούλιο θα βάλει πρόταση για να συμπεριληφθεί με την ίδια έννοια αλλά διαφορετική διατύπωση το γεγονό ότι η ΜΜΕ θα πρέπει να είναι αυτές που θα υποφελούνται κυρίως από την ε, ενεργειακή αποδοτικότητα. Αλλά υπάρχει και η συμφωνία της Natura 2000 μεταξύ των τριών πλευρών. Το πραγματικό πρόβλημα που είχαμε, όπω ανέφερα και προηγουμένω, ήταν το γεγονό ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο ήταν αντίθετοι με την τροπολογία που προτεραιότητα επενδύσεων για την ε, ενεργειακή απόδοση και την δημιουργία ε, και την διανομή ε, ηλεκτρικής ενέργειας μέσω τέτοιου επενδύσεων. Αυτό είναι κάτι με το οποίο διαφωνούμε, διότι θα θέλαμε να υπάρχουν στα πλαίσια των προτεραιοτήτων επενδύσεων ε, σχέδια για να θερμαίνεται με να θερμαίνονται με κοινό τρόπο ολόκληρες περιοχές. Όλοι υπεστήριξαν αυτή την ιδέα, εκτός των δύο εταίρων μας, θα ήθελα να επιμείνουμε εμείς και κάτι άλλο που ε, πάντες δέχθηκαν είναι να έχουμε τις ίδιες διατάξεις στο ERDF, δηλαδή στο ΕΤΠΑ και στο Ταμείο Συνοχής, όταν ασχολούμαστε με προβλήματα ε, απόδοσης ενέργειας για στέγαση ε, και ε, κοινού σχεδίου θέρμανσης κάποιων περιοχών και εργοστάσια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Το Συμβούλιο ήταν αντίθετο με τη ιδέα της ε, θέρμανσης μιας ολόκληρης περιοχής Καταρχάς, σιγά σιγά άλλαξαν θέση ακούγοντα τα διάφορα επιχειρήματα. Ελπίζω λοιπόν ότι τελικά θα αλλάξουν τα πράγματα. Για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και η θέση μας απόλυτα σαφής και ελπίζω ότι θα αλλάξουν τελικά θέση. Τώρα, σε σχέση με αυτά που είπατε Βίκτορ, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονό ότι όταν τα κράτη-μέλη ξέρουν ποια είναι τα συνολικά κονδύλια που διαθέτουν τον Φεβρουάριο ή τον ε, Μάρτιο, θα αρχίσουν να κάνουν αξιολόγηση προτεραιοτήτων και ίσως θα έχουμε και για κάποια ε, τέτοιου είδους θέματα αλλαγή θέσεων. Γιάννη τώρα, όσον αφορά τις ε, μεταβατικές περιόδους, ας με διορθώσει ο Νίκος. Αν θυμάμαι, υπήρχαν κάποιες περιοχές εντός ε, παρενθέσεων εξαφανίστηκε για τον ορισμό αυτών των περιοχών. Υπάρχουν σχόλια για τον Βίκτορ, ο Ιβανς. Μια ερώτηση. Ποιος, πού είναι, στο προσάρτημα θα έχετε τον κατάλογο των σχεδίων. Ποιος ε, αποφασίζει. Εάν λάβει χώρα αυτό το Euro Facility, τι θα γίνει με τον κατάλογο. Δεν ε, ε, θα συμπεριληφθεί αυτός ο κατάλογος στο Ταμείο Συνοχής. Ο καθένας θα έχει το δικό του κατάλογο σχεδίων. Αυτή ήταν η αρχική πρόταση της Επιτροπής. Δεν έχει λόγο ύπαρξης εδώ αυτός ο κατάλογος. Συγγνώμη, μία τελική παρατήρηση. Η Γραμματεία έχει προετοιμάσει πιο λεπτομεριακά τα συμπεράσματα τα οποία καταλήξαμε μετά την τελευταία συνεδρίαση του τριμερού διαλόγου. Την έχετε Χθε το βράδυ υπήρχαμε και μια, μια συνεδρίαση με την ε, Ιρλανδική Προεδρία που ανέλαβε δεσμεύσεις όλη η διαδικασία αυτή να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της δικής τους Προεδρίας. Ίσως λοιπόν τον Φεβρουάριο-τον Μάρτιο θα πρέπει να ψηφίσουμε εμείς ε, έχοντας κατά νου ότι θα είναι έτοιμο το κατά 90, 80-90% το περιεχόμενο των κανονισμών που θέλουμε να ψηφίσουμε τον μαρτιο θα πρεπει να ψηφισουμε εμεις εχοντας κατα νου οτι θα ειναι ετοιμο το κατα 90 80 90 το των κανονισμων που θελουμε να ψηφισουμε το προτασουμε Και αν δεν υπάρχουν άλλα θέματα, θα ήθελα να κλείσω αυτό το θέμα και να σας ενημερώσω ότι η επόμενη συνεδρίαση προβλέπεται για ε, μια μισή ολόκληρη μέρα, 23-24 Ιανουαρίου. Θα έχουμε πολλή δουλειά. Θα έχουμε και την ε, Ιρλανδική Προεδρία. Παρακαλώ, λοιπόν, επειδή θα έχουμε φόρτο εργασία, να είστε όλοι παρόντε. Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο νέο χρόνο εύχομαι σε όλου. Ευχαριστώ και στου διερμηνείς και οι διερμηνεί ευχαριστούν την Πρόεδρο.